And first uh, Το θέμα λοιπόν ε, το απόγευμα είναι η κατάσταση στον τριμερή διάλογο όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ε, ανάπτυξης. Και εδώ πέρα έχουμε τον άνθρωπο κλειδί τον εισηγητή, τον κύριο Πάσκου. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Ουσιαστικά το Συμβούλιο δεν έχει εντολή. Σήμερα συνεδριάζει η Κορεπέρ και ελπίζουν να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να παίξουν κι αυτοί. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το δούμε στις 3 ε, ε, Μαΐου όταν θα έχουμε πάλι τον ε, τριμερή διάλογο αλλά δεν αποκλείεται να χρειαστεί και τέταρτη συνεδρίαση κάπου στο τέλος Μαΐου. Ουσιαστικά αυτά. think. Uh, Mr. Stetina first. Πρώτος ο κύριος Στέτινα. Και μετά ο κύριος Δρογεύσκη. Μετά τον κύριο Στέτινα. Uh, okay, <laughs> thank you. That's, thank you, colleague. Pan poseł Zdrojewski. Ο κύριος Δρογεύσκη, λοιπόν. Βεβαίως, προβληματιζόμαστε προβληματιζόμαστε λόγω της διαδικασίας που παρατείνεται και προσευχόμαστε για τον κύριο Πάσκου. Ελπίζουμε να πετύχει και να μπορέσει να ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια. Όμως, σε αυτό το στάδιο, ουδέν σχόλιον. Θέλω να εκφράσω ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείτε, διότι είναι σημαντικότατη έκθεση. Θέλετε να πείτε κάτι? να ολοκληρώσετε αυτό το θέμα ή να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν αναμονή πρόοδου στον τριμερή διάλογο τελούμε. Παρακαλώ τη γραμματεία να κάνει μια αναδιάταξη εδώ. Περιμένουμε τα μέλη του πάνελ για να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Colleagues, uh, please be patient. We have to, to wait a little Λίγη υπομονή να περιμένουμε λίγο για να τακτοποιηθούμε. So, once more we... Λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, της απογευματινής μαζί με τις διάφορες επιτροπές, τις αρμόδιες, Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις σχέσεις με την Αρμενία, το Ατζερμπαϊτζάν και για τις σύνδεσεις, συμφωνίες σύνδεσης με τη Γεωργία και είναι προνόμιό μου να καλωσορίζω τα διακεκριμένα μέλη του πάνελ για σήμερα εξεβονίμων. Κύριος Λόρενς Μέρεντιθ, διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως ΝΙΕΡ, που είναι υπεύθυνη για τις, ε, σχέσεις με τις χώρες ανατολικής γειτονίας. Ο κ. Ντέρκ Λόρενς, που είναι τμήματάρχης ε, για τις διμερείς σχέσεις με τις χώρες εταιρικής σχέσης, με τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ασίας με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως και μόνη η κυρία, μέλος του πάνελ, τη γνωρίζετε καλά, η κυρία Μάντα Πολ, ερευνήτρια, αναλήτρια για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής του κέντρου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις πολιτικές μελέτες και τέλος γνωστός ο κύριος Ηρακλή Ποκίτζε, αντιπρόεδρος του Γεωργιανού Ινστιτούτου Στατηγικών Μελετών. Και ήταν και στο διπλωματικό σώμα της Γεωργίας στην προηγούμενη καριέρα του. Το θέμα. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο Νότιο Κάφκασο. Εστιαζόμεθα ιδιαίτερα ε, όσον αφορά την ασφάλεια στην Γεωργία θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Μέρεντιθ και μετά στον κύριο Ντέρκ Λόρενς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο, ένα-δύο λεπτά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ. Με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Θα ξεκινήσω περιγράφοντας το όλο σκηνικό. Όταν είπα ότι εκπρόσωπος και επίτροπος ο κ. Χάν ζήτησαν να αναθεωρηθεί η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είχα το προνόμιο να βοηθήσω την προετοιμασία αυτή τη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένας από σημαντικούς λόγους για του οποίου θεώρησαν οι Επίτροποι ότι πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική γειτονία εκ νέου ήταν για να λάβουμε υπόψη τι λίγε εξελίξει και τι αλλαγέ που λαμβάνουν χώρα. Υπήρξε επιθυμία από τις χώρες εταίρους και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Και αυτό διαφάνει στα πρώτα έγγραφα για την εξωτερική πολιτική. Εκεί που έγινε ευρεία δημόσια διαβούλευση. Συμμετείχε και το Κοινοβούλιο, αλλά και κράτη-μέλη και άλλοι εταίροι και διάφορες ομάδες προβληματισμού. Και εκεί είδαμε εκ νέου πόσο σημαντικό θα ήταν στην αναθεωρημένη πολιτική να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ασφάλεια και να βοηθήσουμε τις χώρες εταίρους να γίνουν πιο ανθεκτικές όσον αφορά τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Και βασιζόμενοι επί των πολιτικών στόχων αυτών, εργαστήκαμε άοκνα από, το, από την αναθεώρηση του 2015 του Νοεμβρίου και έγινε κορυφής Ανατολικής Γειτονίας το Νοέμβριο Εκεί συμφώνησαν όλοι επί τεσσάρων προτεραιοτήτων. Το ένα είναι η διακυβέρνηση και η ασφάλεια. Ένα από τα θέματα. Και βάλαμε 20 στόχους για το 2020, ε, θεματολόγοι που στηρίζουν και οι χώρες εταίροι και τα κράτη-μέλη και έχουμε 12 στόχου που να πετύχουμε. Εστιαζόμαστε κυρίως επί τη ασφαλεία σε αυτό το τομέα και ο Ντέρκ Λόρεν από πλευρά τη Υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων θα αναφερθεί εκτενέστερα και λεπτομερέστερα. Ε, στην Ανατολική Γειτονία έχουμε το θέμα των συγκρούσεων. Πέντε από τι έξι χώρε προβληματίζονται από αυτό. Εστιαστήκαμε επί τη Γεωργία και του Νοτιού Καυκάσου. Αρχές εβδομάδας διοργάνωση υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω, σημαντικότατο σεμινάριο εκεί εξετάστηκαν οι συγκρούσεις, συμμετείχαν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και ετοιμάζουμε και οργανώνουμε διάφορα σεμινάρια, διότι κατανοήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συντονισμένοι και τα θεσμικά όργανα να είναι συντονισμένα και να ακούσουμε και κάποιους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, διότι είναι πολύ ευαίσθητα θέματα πλευράς πολιτικής και πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη κατανόηση, με μεγάλη ευαισθησία και θα έλεγα ότι στις διμερείς σχέσεις Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι Γεωργιανοί ε, θέλησαν να τονίσουν ιδιαίτερα τα θέματα ασφαλείας και συμφώνησαν ότι θα πρέπει να διεξαχθεί διάλογος σε υψηλό επίπεδο για θέματα ασφαλείας. Διάλογος Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι μια έξοχη πρωτοβουλία. Συμφώνησαν ε, ο Πρωθυπουργό Γεωργίας και είπατε εκπρόσωπος προ 18 μήνου και ήδη ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και βέβαια αυτή είναι, αυτές οι συζητήσεις εξάγονται σε αυτό, είναι το υψηλότερο επίπεδο συζητήσεων. Συζητάμε όχι μόνο συγκρούσεις αλλά όλες τις απειλές κατά της ασφαλείας. Εγώ προσωπικά μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω και με τον ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι γίνεται, ποιο τμήμα του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα χρησιμοποιηθεί από πλευρά διμερών σχέσεων και περιφερειακών κονδυλίων Συγγνώμη μπαίνω σε τεχνικέ λεπτομέρειε, αλλά είναι αρκετά σημαντικό το θέμα, διότι στον διμερή προπολογισμό αυτά θα πρέπει να του δώσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ε, κυβερνήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα, είναι πιο light η προσέγγιση ε, και είναι θέμα διάθρωση υποστήριξη. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα, ακροθυγώ να αναφερθώ σε δύο διαφορετικά θέματα. Υποστήριξή μα στα πλαίσια των συγκρούσεων θα πρέπει να ελέγχεται από την ύπατη εκπρόσωπο και την εξωτερική δράση δράσης από πλευρά πολιτικής, αλλά πρέπει να έχουμε ευελιξία και επάρκεια στον αφορά τη μέθοδο υποστήριξης με άλλε περιοχές, στα Δυτικά Βαλκάνια. Είδαμε την εμπειρία ότι τα χρήματα σε μια φάση διαμεσολάβησης και διαπραγματεύση αλλάζει τη δυναμική των συζητήσεων. Και να φτάσει καν στη διαδικασία και μετά να σκεφτεί τα χρήματα είναι λιγότερο αποτελεσματικό σαν μέθοδο. Απαιτεί κάποια κατανόηση από το Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη για την ευελιξία που απαιτείται και πώ λειτουργούμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση και το είδο τη υποστήριξη που θέλει να παράσχει κάποιο, διαφέρει. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά την υγεία, την παιδεία, πίν θέματα που μπορεί να, να φανούν. Uh, Παραδείγματο χάρη πω ε, κάποια ζυζάνια μπορεί να πειράσουν κάποια σοδιά. Παραδείγματο χάρη σε περίπτωση προβλήματο μπορούμε να δώσουμε κάποια βοήθεια που είναι κάτι κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη περιοχή, αλλά δεν είναι πολιτικά τόσο σημαντικό. Και δεν θα το προβλέπαμε πριν προκύψει η κρίση ότι χρειαζόταν αυτή την υποστήριξη. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Λοιπόν, χρειάζεται ευελιξία και υποστήριξη. Είναι μου σημασία σε αυτό. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω. Αλλά πιστεύω και θεωρώ ότι στον προγραμματισμό χρειάζεται ευαισθησία όσον αφορά τα προβλήματα και τις συγκρούσεις. Διότι και στις χώρες του Καυκάσου ε, είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Και όποια χρήματα δαπανούν αυτές οι τρεις κυβερνήσεις για ασφάλεια, για άμυνα. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους τομείς, όπως για την υγεία και την παιδεία. Βλέπετε έχουν αυστηρά ε, δημοσιονομικά πλαίσια. Άλλαξε η προσέγγιση όσον αφορά τι παγωμένε σειράξει στη Σύνοδο Κορυφή. Δεν είναι παγωμένε, είναι παρατεταμένε οι κρίσει και συγκρούσει, θα έλεγα. Οι ηγέτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω και εταίροι συμφώνησαν επί και θα λένε τώρα ανεπίλητε συγκρούσει. Άλλαξε η διατύπωση. Αντί παγωμένε, ανεπίλητε. Πολύ σύντομα λοιπόν. Είναι ευρύτερο κεφάλαιο η σύγκρουση, ε, η ασφάλεια μάλλον. Καλύπτει πολλά για τη Γεωργία. Όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων των ταξιδιωτικών και το διάλογο, οι πολίτες της Γεωργίας ανέλαβαν υποχρεώσεις για την ασφάλεια, για το οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών. Πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κατσαπλιάδες οι οποίοι τελικά διακινούν αυτά τα ναρκωτικά. Λοιπόν, και θα πρέπει να παράσχουμε υποστήριξη προσπάθειας που καταβάλουν και από την πλευρά μου προσπάθησα να κινηθώ και σε άλλα πλαίσια, στον κυβερνοχώρο, παραπληροφόρηση που είναι μεγάλα προβλήματα. Και όχι μόνο στη Γεωργία, σε όλη την περιοχή. Και μαζί με τη Stratcom, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα εξετάσαμε αυτά. Τι θετικά μηνύματα που να στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια πρακτικά θέματα πρέπει να διαθετηθούν. Και θα σταματήσω εδώ γιατί έχουμε και άλλα μέρη του πάνω που αναφερθούν σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Ντίκ Λόρενς από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια και ο Λόρενς μας έκανε μια καλή επισκόπηση του γενικού πλαισίου και της πολιτικής, τότε εγώ θα μπω κατευθείαν στο θέμα της ασφάλειας ε, στη Γεωργία, που είναι και το βασικό θέμα της σημερινής μας ε, συνάντησης. Η, η Ο χάρτης και η ασφάλεια, ε, το θέμα της ασφάλειας είναι σε καλή κατάσταση αλλά ευάλωτη. Μετά τις εχθροπραξίες το 2008 υπήρξαν κάποιες εξελίξεις περάσαμε σε παρατεταμένη ή ανεπίλητη σύγκρουση. Ε, τώρα η κατάσταση δεν είναι τόσο οξία. Η, σύγκρουση ουσιαστικά λόγω της δυναμικής, της δυναμικής ε, στην πραγματικότητα έχει παγιωθεί. Ε, οι σχέσεις Γεωργίας και Ρωσίας, Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν βελτιωθεί ε, σε περιοχές ε, όπως τουρισμός, μεταφορές και εμπόριο που δεν έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση. Υπάρχουν όμως το 2017 ε, υπήρχαν προβλήματα. Η πρόοδος σε ορισμένους τομείς όμως δεν ε, επηρέασε τον χώρο της ασφάλειας. Οι επίσημες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας δεν έχουν αποκατασταθεί. Οι προϋποθέσεις ε, από πλευράς Γεωργίας είναι ότι θα πρέπει η Ρωσική Ομοσπονδία να μην αναγνωρίσει πια την ανεξαρτησία των περιοχών που έχουν φύγει και να, φύγει, να φύγουν τα στρατεύματα τα οποία βρίσκονται εκεί, τα ρωσικά στρατεύματα. Τώρα, για τις δύο περιοχές που έχουν προχωρήσει, η Απχασία και Νότια Οσετία ε, βρίσκονται υπό την εμπειρία, ακόμα πιο έντονη εμπειρία της Ρωσίας μέσω νομικών, πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών ε, και εκπαιδευτικών μέτρων καθώς και πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου. Αυτά τα είπε και ο Διευθυντή. Ω αποτέλεσμα, ο διαχωρισμό ανάμεσα στην, στο διοικητικό, ε, διοικητική περιφέρεια του, της Τυφλίδας και τις περιοχές αυτές έχει αυξηθεί. Ε, και θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να μετασχηματιστεί η σύγκρουση α, βραχ, και για να επιληθεί βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα είναι οι μικρές πιθανότητες. Μια νέα φάση, έχει, μάλλον έχει ξεκινήσει αυτό, αυτή το 2017, που οδήγησε σε αναβάθμιση των, του εξοπλισμού. Έκλεισαν κάποια περάσματα διέλευσης, πιο έντονη, έντονη αστυνόμευση, πιο αυτή περιορισμοί σε ό,τι αφορά τα έγγραφα και όσοι χρησιμοποιούν ανεπίσημα σημεία διέλευσης τιμωρούνται. Επομένως, οι διοικητικές ε, συνοριακές γραμμές ε, έχουν γίνει ακόμα πιο απαραβίαστες, περιορίζοντας το, περι... το περιθώριο ελευθερίας του τοπικού πληθυσμού. Φυσικά, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέμα, το θέμα της ε, EUAM, της αποστολής δηλαδή παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου που είναι και η μόνη αποστολή στην περιοχή. Εφαρμόζει την εντολή της στην διοικητική επικράτεια της Τυφλίδας, αλλά δυστυχώς δεν έχει πρόσβαση στις ε, περιοχές που έχουν αποχωρήσει και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση με τα έξι σημεία ε, της η Αυγούστου του 2008, τα, σημεία που συμφωνήθηκαν και τα μέτρα ε, που συμφωνήθηκαν εν συνεχεία το Σεπτέμβριο του 2008. Πέρα από την UMM έχουμε και την τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίζει το ρόλο του διευκολυντή και διαμεσολαβητή των δύο μερών και είναι συμπρόεδρος στην, ε, στις διεθνείς συζητήσεις της Γενέβης. Πιστεύουμε ότι μια ουσιαστική αλλαγή τη δυναμική τη σύγκρουση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο για γίνουν σοβαρέ πολιτικέ αλλαγέ, περισσότερε δημοκρατικέ και οικονομικέ εξελίξει και μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη ανάμεσα στο Τουκούμι και, στο Τσικάμπι και, στο, και στην Τυφλίδα. λέει το Σοχούμι. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και να συνεισφέρουν και διεθνεί παράγοντε. Η Γεωργία παίζει σημαντικό ρόλο ε, και είναι σημαντικό να συνεχίζει την προσπάθεια μετασχηματισμού ή επίλυση της σύγκρουσης. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και σε μια συντονισμένη εθνική στρατηγική και να συνοδευτεί από μια ε, ανακοίνωση και ενημέρωση του πληθυσμού της Γεωργίας ε, ότι υπάρχει τάση προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι το πρόσφατο πακέτο πρωτοβουλειών που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση της Γεωργίας είναι ένα σημαντικό βήμα. Αυτά τα μέτρα μπορούν να είναι υποφελή για τους πολίτες που ζουν και στις δύο πλευρές της, ε, του συνοριακού, της συνοριακής γραμμής ε, και το εμπόριο, η κινητικότητα και η εκπαίδευση μπορούν να υποφεληθούν. Ε, οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται σε επαφή με τις περιοχές της Γεωργίας, με πρωτοβουλίες για να υπάρξουν γέφυρες ανάμεσα στις δύο πλευρές και με την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων βοηθάει ε, και αυτή. Τώρα, ποια είναι η συνεισφορά ε, της ε, Γεωργίας στην ΚΠΑ και ποια είναι η συνεργασία ανάμεσα στη Γεωργία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα θέματα ασφάλειας. Η Γεωργία σύν τον χρόνο έχει δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αυτή τη στιγμή συνεισφέρει σε δύο στολές ε, στη EUTRMCA ε, Φεβρουάριο του 2017 με 35.000 ε, στρατιώτες και στο Μαλί με έναν αξιωματικό από τον Ιανουάριο του 2016. Επιπλέον, ε, διαβουλεύσεις προσωπικού και συμμετοχή σε δραστηριότητες εκπαίδευσης είναι τμήμα της συνεργασίας Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, κάτι που υπόθηκε ήδη, έχουμε ένα νέο εργαλείο που είναι ο άτυπο στρατηγικό διάλογος για την ασφάλεια. Ο πρώτος έγινε στο, στη τον Οκτώβριο του 2017 και η Γεωργία εξέφρασε τότε το ενδιαφέρον να ενισχύσει την συνεργασία για την ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως υπό τη μορφή οικοδόμηση δυναμικού στους τομεί τη προστασία των αμάχων, αντιμετώπιση των επιγόντων ε, ειδικά μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές, ε, προστασία των συνόρων και σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας. Ε, η Γεωργία επίσης έχει και πολλές ιδέες και πολλές πρωτοβουλίες για το πώς θα προχωρήσει αυτός ο διάλογος και η συνεργασία. Δεν θα μιλήσω για την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν τώρα, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις για αυτές τις δύο χώρες θα τις απαντήσω. Στο βαθμό που μπορώ φυσικά. Σας ευχαριστώ κύριε Λόρεντς. Τώρα έχουμε δύο ειδικού ε, εγνωσμένου κύριους. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μανταπόλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και είμαι και φίλη της Γεωργίας. Ε, ειλικρινά μιλώντας, δεν ήταν πολύ τυχερή η Γεωργία από πλευράς γεωγραφίας, αλλά θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα, γιατί αν ήταν λίγο πιο δυτικά, ας πούμε στα Δυτικά Βαλκάνια, θα ήταν ήδη υποψήφια χώρα και θα ήταν ήδη μέλος του ΝΑΤΟ. Τραγικό λοιπόν αυτό, γιατί ο Νότιος Κάφκασος είναι μια πολύ στρατιωτικοποιημένη και επικίνδυνη περιοχή από τις χειρότερες στον κόσμο Δέκα σημεία έχω να αναφέρω, θα είμαι σύντομη όμως και ζητώ συγγνώμη αν ξεπεράσω τον χρόνο. Πρώτον, έχουμε την ρωσική κατοχή. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι το 20% της χώρας εξακολουθεί να κατέχεται από την Ρωσία και αυτό είναι το οξύτερο πρόβλημα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα. Από το 2008 που είχαμε τον πόλεμο η Ρωσία έχει αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία και στην Νότια Οσετία και στην Απχασία. Ουσιαστικά και οι δύο περιοχές εξαρτώνται πλέον από την Ρωσία και η Ρωσία ελέγχει τα πάντα. Υπάρχουν χιλιάδες ε, Ρώσοι στρατιώτες και οπλισμός στις δύο περιοχές και οι κατεχόμενες περιοχές είναι πολύ χρήσιμες ε, στους Ρώσους γιατί από εκεί προβάλλουν ισχύ σε ολόκληρη την ε, περιοχή και δημιουργούν αστάθεια ε, όταν το κρίνουν ε, χρήσιμο και βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις συγκρούσεις. Δεύτερον, έχουμε τις τεράστιες στρατιωτικές ασχήσεις που διεξάγει η Ρωσία. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση των υπηρεσιών ασφαλείας της Γεωργίας, μόνο το 2017 η Ρωσία διεξήγει πάνω από 100 παράνομες ε, στρατιωτικές ασκήσεις στα κατεχόμενα. Η τελευταία ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν μια τεράστια άσκηση που καλύπτει την Νότια Ρωσία, την κατεχόμενη Κρυμαία, την Αυχαζία και την Νότια Οσετία. Περιλάμβανε 8.000 στρατιώτες ε, και εξοπλισμό. Ε, ρουκέτες, πυροβολικό κτλ. Έτσι λοιπόν τίθεται σε κίνδυνο όχι μόνο η Γεωργία αλλά ολόκληρος ο Νότιος Καύκασος είναι ένας τεράστιος κίνδυνος ασφαλείας αλλά και για τις υποδομές, το σιδηρόδρομο, τους αγωγούς που πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Το ανέφερε. ο Επίσης, το επόμενο θέμα έχουμε το ειρηνευτικό σχέδιο των έξι σημείων, το οποίο δεν εφαρμόζει η Ρωσία καθόλου. Το πρώτο σημείο είναι ότι πρέπει να αποσυρθούν οι ρωσικές δυνάμεις ε, στην γραμμή που ήταν πριν από το 2008 και το δεύτερο βεβαίω αφορά ελεύθερη πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια. Ούτε αυτό γίνεται. Και βεβαίω αναφερθήκαμε ήδη στην πρόσβαση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρώτησα λοιπόν ποιες είναι οι συνέπειες της ε, μη εφαρμογής ε, και δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Και το τέταρτο είναι βεβαίως ε, η διακριτική μεταχείριση στους γεωργιανούς που ζουν στα κατεχόμενα, παράνομη κράτηση, απαγωγές στο λεγόμενο σύνορο. Μία από τις τελευταίες περιπτώσεις που μάλλον θα έχετε ακούσει ήταν ο Αχιλέας τα Βίλη που πέθανε υποκράτηση στις 23 ε, Φεβρουαρίου υπό περίεργες συνθήκες. Ποιες είναι οι συνέπειες και πάλι καμία. Και πάλι το θέμα της συνοριοποίησης. Τι συνέπειες έχει και αυτό. Πάλι καμία συνέπεια. Σημείο 6. Ο υβριδικός πόλεμος, η παραπληροφόρηση, οι κυβερνοεπιθέσεις που είναι μια σημαντική απειλή ασφαλείας. Ε, ούτε και αυτό είναι καινούριο για την Γεωργία γιατί η Γεωργία το αντιμετωπίζει αυτό εδώ και χρόνια πριν ε, απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βεβαίως έχει αυξηθεί μετά από τον πόλεμο του 2008 σημείο 7 Έχουμε τη στρατιωτικοποίηση της Μαύρης Θάλασσας που επίσης αποτελεί απειλή για την Γεωργία και την ευρύτερη περιοχή. Η Γεωργία βρέχεται από την Μαύρη Θάλασσα και έχει ενταθεί αυτή η στρατιωτικοποίηση από την παράνομη ένταξη ε, με συγχωρείτε, προσάρτηση της ε, Κρυμαίας, ε, η οποία είναι μια τεράστια στρατιωτική βάση και χρησιμοποιείται και για την Συρία και έχει ενταχθεί στο ρωσικό σύστημα με τις βάσεις στην Αρμενία και αλλού και στο Ροστόφ επίσης. Όγδο έχουμε την σύγκριση του Ναγκόρνο Καραμπάχ και εκεί πέρα έχουμε μια απειλή για την ασφάλεια της Γεωργίας όχι μόνο λόγω των ε, παραβιάσεων της ε, κατάπαυσης ε, του πυρός που όπως είδαμε οδήγησαν και σε ένα πόλεμο τεσσάρων ημερών στο παρελθόν και να έχουμε αναζωπήρωση δηλαδή του πολέμου αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν αλλά όλες τις χώρες της περιοχής και τις υποδομές και θα ανοίξει την πόρτα για να έρθουν πιθανώς και ρώσικα ειρηνευτικά στρατεύματα. Και έτσι μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ α, της αζερικής και αρμενικής κοινότητας ε, που ζουν στην Γεωργία. Να σας ε, αυτό δεν έχει σχέση βεβαίως με τους ε, Ρώσους, αυτό που θα πω, αλλά είναι οι οικονομικές και οι κοινωνικές προκλήσεις. Έχει μεγάλη σημασία η οικονομική ανάπτυξη για την εθνική ασφάλεια γιατί βεβαίως ε, πρέπει να δημιουργηθούν και ισχυροί θεσμοί και νομίζω ότι έχουμε μια θετική θα έλεγα δυναμική στην γεωργία για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να καταπολεμηθεί η διαφθορά να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη η ανταγωνιστικότητα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για να μειωθεί η ανεργία. Γιατί η ανεργία μπορεί να δημιουργήσει και άλλες εντάσεις και βεβαίως να ενισχυθεί και η ενεργειακή ασφάλεια. Και τέλος, κάτι το οποίο αφορά τις διαδικασίες ευρωατλαντικής ένταξης που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να ενισχυθεί η αντοχή της χώρας Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη έναν οδικό χάρτη για μεταρρυθμίσεις και παίζει ένα σημαντικό ρόλο μέσω της αποστολής της στην Γεωργία και συμπροεδρεύει και στις ε, συζητήσεις ε, στην Γενέβη οι οποίες βεβαίως κάπου έχουν κολλήσει, αν μου επιτρέπετε, ε, διπλωματικά να το εκφράσω. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε το status quo. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερη δημιουργικότητα για να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις. Και τέλος, η σχέση της Γεωργίας με το ΝΑΤΟ. Είναι νομίζω πολύ στενή. Το ΝΑΤΟ έχει βοηθήσει να μετασχηματιστεί ο στρατός της Γεωργίας σε έναν δυτικό στρατό και βεβαίως πληρεί τις προτεγραφές του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες σε αντίθεση με πολλά μέλη του ΝΑΤΟ αλλά βεβαίως η ένταξη στο ΝΑΤΟ ακόμα είναι πολύ μακρινή. Ελπίζουμε ότι στην σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ θα έχουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις για να περάσει η σχέση σε ένα άλλο επίπεδο. Και τέλος, δύο σημαντικά βήματα είναι η περιφερειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα που έχει μεγάλη σημασία για την αντοχή της χώρας και στον τομέα της ασφαλείας και στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με σημαντικές χώρες όπως η Κίνα. Βλέπουμε ότι η Γεωργία και η Κίνα έχουν ενισχύσει τις οικονομικές τους σχέσεις και όπως είδαμε παραδείγματος χάρη και με την Τουρκία και υπάρχει και η νέα πρωτοβουλία της ε, κυβέρνησης για τα κατεχόμενα και αυτό ήταν νομίζω κάτι το πολύ θετικό και με συγχωρείτε αν ξεπέρασα το δεκάλεπτο. λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Απόλ. Τέλος. Ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Στατηγικών Μελετών της Γεωργίας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε. Ηράκλειο, τιτάνιο έργο να μιλάει κανείς τελευταίος διότι πολλά ήδη καλύφθηκαν. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Να σας πω γιατί η Ρωσία κινείται του τρόπος και γιατί έχει θέσει αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Η ασφάλεια επιτόπου, πρώτο θέμα. Η Ρωσία έχει περίπου 5.000 στρατιωτικούς σε κάθε κατεχόμενη περιοχή. Να πούμε ότι έχει βάλει κίνηση στις μονάδες στη νότια περιοχή. Έχει εξυγχρονίσει αυτές τις περιοχές. Δημιουργεί στατιωτικές υποδομές. Και έχει τέτοια διαδικασία διαταγών που ακολουθείται που έχει βελτιώσει την οργάνωση και τις γραμμές επικοινωνιών. Έχει και τους μεθοριοφύλακες, FSS όπως αποκαλούνται, τους ίδιους χρησιμοποιεί και αλλού τους μεθοριοφύλακες αυτούς. Σ' άλλα σύνορά τη. Περίπου 13.000 μεθοριοφύλακες χρησιμοποιεί. 13.000 λοιπόν στατιωτικούς και FSS έχουμε επιτόπου, συνολικά. Σοβαρό πρόβλημα. Να αναφερθώ και στην ανάπτυξη επιτοπίων υποδομών. Συνεχώς βελτιώνουν τις υποδομές. Και η ρωσική παρουσία δεν αφορά μόνο την προβολή ισχύω εντός της Γεωργίας, διότι βλέποντας τον εξοπλισμό, το είδος του εξοπλισμού και την ποιότητά του, η προβολή ισχύω έχει στόχο πέρα από τα σύνορα της Γεωργίας, πέρα τον Κάφκασο, τον Εύξηνο Πόντο. Έχει τακτικά πυραυλικά συστήματα, αεράμινα και επιθετικά όπλα και συστήματα. Πέρα από αυτό. Δυνατότητες αναγνώρισης μη επανδρομένα οχήματα αναγνωριστικά, ελικόπτερα. Έχει στατικοποιηθεί η περιοχή και οι δύο περιοχές. Και τα άλλο που αναφέρθηκε. Οι ασκήσεις. Έχουν εντατικοποιηθεί οι ασκήσεις. Σε όλες αυτές τις περιοχές. Αυτές που συζητούμε. Συνεχής η τάση αυτή τα τελευταία. Το 2018 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Βέβαια, πρέπει να μιλήσουμε και για τις κρατήσεις. Το 2017, 178 φυλακίσεις υπήρξαν. Φέτος, 13 σε κάθε περιοχή από τις κατεχόμενες. Εξακολουθεί να είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό για τον τόπιο πληθυσμό της Γεωργίας αλλά και την κυβέρνηση της Τυφλίδας. Του Τατουνασφίλη την υπόθεση τη συνδέω ε, μαζί με αυτό, διότι ο Τατουνασβίλη, πολίτης της Γεωργίας, απήχθη στο Χαλγκόρι, την κατεχόμενη περιοχή, περίπου 1,5 μήνα πριν. Και σε μία μέρα βρέθηκε νεκρός. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Για τον επόμενο μήνα οι Ρώσοι και άλλες μονάδες επιτόπου δεν παρέδωσαν ε, τη σωρό. Προσπάθησαν να συγκαλύψουν τα βασανιστήρια που υπέστη. Τι σουλές, τα σημάδια. Άλλα σημάδια στη σωρό του, του ασβίλη. Τα εκάλυψαν. Παρεδόθηκε η σωρός του ένα μήνα αργότερα μετά τη σύλληψη και κράτησή του. Συνεχίζεται η ατιμορρησία. Και έχουμε και τη δολοφονία του Τροζόρια που έγινε σε αυτή την περιοχή, στα σύνορα με την κατεχόμενη Απκασία. Ατιμορρησία και εσύ. Οι έρευνες και των δύο υποθέσεων δεν διεξήχθησαν επισήμως τουλάχιστον. Δεν έχουν διαλευκανθεί υποθέσεις. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Επικρατεί ένας εκροσισμός στις περιοχές. Και οι πρεσβείες επιτόπιες δίνουν διαβατήρια, εκδίδουν παράνομα διαβατήρια στον τόπιο πληθυσμό και είναι και το γλωσσικό στοιχείο της κατοχής. Προφανέστατο. Όσον αφορά τη διδασκαλία στα σχολεία, την παιδεία, στην τοπική γλώσσα, στην Απκαζία, το πρόβλημα σχετιζόταν με την αφαίρεση ε, της γλώσσας της Γεωργίας, της Γεωργιανής, όσον αφορά ε, γλώσσα εκμάθησης διδασκαλίας. Σταδιακά, βγάζουν τη γεωργιανή γλώσσα από πρώτη με πέμπτη τάξη. Και συνεχώς αφαιρείται από κάθε τάξη που ακολουθεί η δασκαλία σε αυτή τη γλώσσα. Όλοι οι Γεωργιανοί τελικά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν, να σπουδάσουν στη γλώσσα τους. Θα λησμονηθεί η γλώσσα. Εκροσισμός επικρατεί. Η Ρωσία επενδύει μεγάλα ποσά γι' αυτό. Μέσω των ΜΚΙ όπως αποκαλούνται και μέσω της παροχής ε, διδακτικού προσωπικού. Η Ρωσία λοιπόν εκμεταλλεύεται την αδυναμία παροχής ε, κάλυψης των θέσεων διδασκαλίας και παρέχει τους δικούς διδασκάλους που διδάσκουν κυρίως τα ρωσικά. Έχουμε και απρόβλεπτες εξελίξεις. Καμιά φορά εβδομαδιαία καθημερινά συμβαίνουν απρόβλεπτα. Λοιπόν, πώς βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί κινείται με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία. Σωστά υπόθηκε ότι είναι εύθραυστη η κατάσταση. Ε, έχει όλα τα μέσα η Ρωσία. Στρατό, δυνάμεις, εξοπλισμό στατιωτικό. Και έχει αρπάξει στα νύχια τη στρατηγικά τη Γεωργία. Ε, και έχει και στα χέρια της τον αυτοκινητόδρομο προς την Τυφλίδα. Άρα ε, υπάρχει έλλειψη προβλεψιμότητας όσον αφορά την καθημερινή ζωή στη Γεωργία. Παρ' όλα αυτά εξελίσσεται η Γεωργία. Για τη Ρωσία είναι μη γραμμική η μάχη που δίνει, προσπάθεια που καταβάλει. Δεν εστιαζόμεθα μόνο στα σοβαρά επεισόδια από το 2008, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία κινείται και ασκεί τις πολεμικές επιχειρήσεις επιτόπου. Τέσσερι παράγοντες χαρακτηρίζουν την προσπάθειά της. Αυτού του είδους οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν συνεχή φύση. Ας αφήσει η κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Όλοι το αισθάνονται ότι κάτι τρέχει αλλά έχει διαφορετικό νόημα. Συνδυάζει συμβατικά και μη συμβατικά μέσα και μεθόδους. Το συζητήσαμε εκτενώς και προηγουμένως. Βασίζεται σε φορείς κρατικούς και μη κρατικούς. Και στη Γεωργία και στην Ουκρανία και αλλού. Τέταρτον, εξίσου σημαντικό, βασίζεται σε μεθόδους ε, προπαγάνδας. Το εφάρμοσε στη Γεωργία. Η Ρωσία έχει πολλούς μυστικούς πράκτορες επιτόπου εντός της Γεωργίας. Έχουν δυσδύσεις στις ΜΚΟ, σε ομάδες προβληματισμού κλπ. Στα ΜΜΕ επηρεάζει τα ΜΜΕ, επηρεάζονται τα μηνύματα που διαβάζονται από τα ΜΜΕ. Γιατί το κάνει αυτό η Ρωσία. Έχει τρεις στρατηγικούς στόχους πιστεύω. Πρώτον, θέλει να επιβάλλει το μονομερές ε, τσάτος κουβό, ε, το ρωσικό επιτόπου, και πέρα από τις άμεσες περιοχές θέλει να υπονομεύσει τους φιλοδυτικούς, τις φιλοδυτικές τάσεις και στη Γεωργία και αλλού. Όχι μόνο η Γεωργία της απασχολεί, αλλά και άλλοι. Θέλει να δώσει το παράδειγμα μέσα της Γεωργίας η Ρωσία. Ότι πρέπει να εφαρμοστούν και να επιτραπούν αυτά που θέλει το Κρεμλίνο και τίποτα άλλο. Και είναι το δόγμα περιορισμένης κυριαρχίας. Σοβιετικό δόγμα ήταν αυτό όταν επικρατούσαν οι σοσιαλιστικέ εποχές, οι κομμουνιστικές εποχές. Αυτό έχει υπόψη τη Ρωσία όταν μιλάμε για την έφταστη κυριαρχία κάθε κράτους που την περιβάλλει. Θέλει να έχει βέτο σε θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τη Ρωσία. α πούμε ασφάλεια ή γενικότερα θέματα. Κατεύθυνση της χώρας Φερρυπίν. Να σταματήσω και με τα χαράς να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και προσωπικά. που αναφερθήκατε σε αυτό το δόγμα για την περιορισμένη κυριαρχία. Μην το ξεχνάμε. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή η συνεδρίαση γίνεται σε συνδυασμό με μια άλλη με μια άλλη επιτροπή, συμμετέχουν και μέλη μια άλλη επιτροπή. Ο πρόεδρο μια άλλη επιτροπή είναι εδώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν δίνοντα το λόγο τον κύριο Καρύμ. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένο στην αίθουσα. Είμαι ε, πρόεδρο τη Επιτροπή του Κώδικα Διοντολογία. Ε, γι' αυτό ακριβώ είχαμε κάποια δουλειά εκεί και καθυστέρησα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σα ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσει σα. Επρόκειτο να κάνω τις αρχικές παρατηρήσεις. Αλλά τώρα απλώς θα κάνω τις καταληκτικές παρατηρήσεις για τις παρουσιάσεις που ήδη έγιναν. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ακρόαση, πρέπει να σας πω ότι ο χρονισμός είναι καταπληκτικός, είναι τέλειος. Γιατί αργότερα, σήμερα, εγώ θα ε, υποδεχθώ ε, τους ομολόγους μας από το Γεωργιανό Κοινοβούλιο που ήρθαν εδώ για την έκτη ε, συνάντηση της ε, Διακοινοβουλευτικής Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, αλλά κυρίως η ασφάλεια στη Γεωργία και στο Νότιο Κάφκασο εν γέννη. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τον Νότιο Κάφκασο παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στις κατεχόμενες περιοχές, οι κάθετος αποσχιστήσεις περιοχές και την ε, κατάσταση και τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαμένουν στις περιοχές αυτές και κοντά στην διοικητική συνοριακή γραμμή. Οι αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι σε αυτές τις ε, κατεχόμενες περιοχές της Απχασίας και Νότιας Οσετίας είναι απλές. Καταρχάς, ε, σεβόμαστε την ε, εδαφική και εθνική κυριαρχία της Γεωργίας με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τη, που σημαίνει πολιτική μη αναγνώρισης. Δεύτερον, είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε σε ειρηνική επίλυση της σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας, συμπεριλαμβάνοντας και τις διεθνείς συζητήσεις της Γενέβης ε, της αποστολής παρακολούθησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Νότιο Κάφκασο και την κρίση της ε, Γεωργίας. Στηρίζουμε την ε, Γεωργία για να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση που κάνουν οι Ρώσοι και τις συνέπειες της σύγκρουσης στις κατεχόμενες περιοχές, να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να ε, μειώσουν τις εντάσεις στις γειτονικέ περιοχές ε, δίπλα από την διοικητική συνοριακή γραμμή. Η αντιπροσωπεία μας κατ' επανάληψη έχει συγχαρεί τις ρωσικές αρχές για τον επικοδομητικό ε, και ρεαλιστικό τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν τους πληθυσμούς των κατεχόμενων περιοχών προς το συμφέρον όλων των πολιτών της Γεωργίας. Αυτή η διάθεση για διάλογο έχει φανεί και πριν από λίγες ε, εβδομάδες που έκανε μια παρουσίαση το Γεωργιανό Κοινοβούλιο για μια πρωτοβουλία για ειρήνη που θα μπορούσε να είναι υποφελής για τους πολίτες που ζουν και από τις δύο μεριές της διαχωριστικής γραμμής ε, προς το καλό του εμπορίου, της κινητικότητας και του και τη εκπαίδευση. Έχουμε ένα πρόγραμμα επίση απελευθέρωση από τις υποχρεώσει θεωρήσεων, ε, πολύ σημαντικό, που επηρεάζει πραγματικά άμεσα αυτές τις κατεχόμενες περιοχές θετικά. Επίσης, ε, με μεγάλη προσοχή προσέξαμε την επίπτωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην περιοχή, γιατί πρέπει να δημιουργηθούν νέα κανάλια μεταξύ των κοινωνιών των δύο που ζουν ε, ένθεν και έθεν της ε, συνοριακής γραμμής για να υλοποιηθεί η συμφωνία και να έχει επιπτώσεις και στους πληθυσμούς. Δηλαδή, η προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ρωσίας, οι στρατηγικές προσάρτησης ε, υπόγειες, καθώς και η διαδικασία ε, συνοριοποίησης, όλα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, όπως φαίνεται και από το πλαδεσιασμό των στρατιωτικών γυμνασίων και ασκήσεων των τελευταίων μηνών ή για την, μέσω της προσ, πρόσφατης απόφασης ε, της ε, Μόσχας να βάλει και νέες δυνάμεις στρατού στις ρωσικές δυνάμεις που είναι επιτόπου. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποτρέψουμε και θα μειώσουμε αυτές τις απειλές και, θα, και να επαναδιατυπώσουμε και να διατρανώσουμε την ε, αλληλεγγύη μας με τη Γεωργία. Θα ήθελα να ξανατονίσω ως Πρόεδρος ότι έχω εκδώσει μια δήλωση για τον τραγικό ε, θάνατο ενός γεωργιανού πολίτη σε κράτηση του Τατούσα Βίλη το Φεβρουάριο του 2018 και ξέρω ότι αναφέρθηκαν και διάφοροι ομιλητές του πάνελ στην, στο θάνατο αυτό. Πολλές από τις συζητήσεις ε, αφορούν την κατάσταση της ασφάλειας στη Γεωργία, όντως. Όμως, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τη σύγκρουση για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ε, το status quo δεν είναι βιώσιμο. Για τρεις δεκαετίες αυτή η σύγκρουση έχει προκαλέσει θάνατο αμάχων και στρατιωτών και έχει παρεμποδίσει την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης περιοχής. Τα μέλη της αποστολής μας ε, εκφράζουν την παρέγκλητη υποστήριξη στις προσπάθειες που κάνουν ε, επιτόπου για να επιληθεί η ειρηνικά η κατάσταση και προς μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης. Αυτές οι προσπάθειες συμπληρώνονται από τη δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθηθεί η εμπιστοσύνη και η ειρήνη ε, μέσω της εφαρμογής της ευρωπαϊκής ιτερικής σχέσης για την ειρηνική διευθέτηση της α, ε, σύγκρουσης στον Αγκόνο Καραπάχ, ούτως ώστε ε, η κοινωνία των πολιτών η Αζέρικη και του Αζερμπαϊτζάν και ε, της Αρμενίας, συγγνώμη, να έρθουν πιο κοντά. Ε, υπάρχει ο κύριος Κλάρκ, ο ειδικός απεσταλμένος και ε, χαιρετίζουμε επίσης την ε, αναγνώριση της Γεωργίας για την αποστολή μας εκεί. Συνεχίζονται οι συζητήσει υψηλού επίπεδου Αρμενία και Αζερβαϊτζάν για να χτιστούν για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνη και ανανέωση του διαλόγου, τόσο ώστε να υπάρχει πιο επικοδομητική ε, πιο επικοδομητικό πλαίσιο για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Τέλος, θα ήθελα, Πρόεδρε, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους τις συστάσεις της 15ης Νοεμβρίου του 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και στην Υπηρεσία εξωτερική δράση για την ε, Ανατολική Γειτονία ε, πριν από την ε, τελευταία σύνοδο. Εκεί ζητάμε από αυτά τα όργανα να επικυρώσουν τις νέες συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κα, καθενός από τα μέρη ε, ως προϋπόθεση για να επιληθεί η σύγκρουση. Νομίζω ότι θα ήταν ένας θαυμάσιος ε, μοχλός πίεσης που έχουμε. Μπαίνουμε τώρα στη δέκατη επέτειο από τη στιγμή που η Ρωσία άρχισε να κατέχει αυτές τις δύο περιοχές, νότιο Νότια Οσετία και Απχασία, θα πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να σκεφτούμε πολύ σοβαρά την περίπτωση ε, να συντάξουμε ένα ψήφισμα για να τιμήσουμε αυτή την επέτειο και ως Πρόεδρος θα υποστηρίξω τη συγγραφή ενός τέτοιου ψηφίσματος για να αναγνωριστεί πια όρος κατεχόμενα εδάφη. Σας ευχαριστώ κύριε πριν ε, δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, να σας ε, ενημερώσω πως ε, σε δύο εβδομάδες η αποστολή μας θα πάει στην Γεωργία όχι μόνο για πολιτικές συζητήσεις στην Τυφλίδα αλλά θα πάμε πιο κοντά στη λεγόμενη γραμμή επαφής στην Αφχαζία αυτή τη φορά στο Ζαγντίντι και αλλού και αναμένουμε αυτή την επίσκεψη και πέντε το λόγο σε άλλους ομιλητές θα ήθελα να παρακαλέσω τους ειδικούς μας να αναφερθούν στις τελευταίες εξελίξεις ε, στην ε, Αρμενία. Ειδικά ε, δεδομένων των διαμαρτυριών και της κοινωνίας των πολιτών που είναι πολύ ζωντανή στην Αρμενία. Και με ενδιαφέρει να μάθω τι άποψη έχετε κι εσείς. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό καμιά φορά να κάνουμε έναν απολογισμό. Και όσον αφορά την κατάσταση στην Γεωργία πρέπει να πούμε ότι αφενός η ρωσική πλευρά ενισχύει ε, τα στρατεύματά της ε, και ναι. Καθιστά εκεί. Υποδομές ε, στα κατεχόμενα. Είχαμε επισκεφτεί επίση εκεί την Ευρωπαϊκή Αποστολή. Είδαμε κάποιες στρατιωτικέ εγκαταστάσεις και έναν ε, τεράστιο δρόμο. Ε, γιατί οι κοιλάδες στην Νότια Οσετία πηγαίνουν από βορρά προς νότον, ενώ έχτισαν έναν τεράστιο δρόμο από Ανατολή προς Δύση που θα κόστησε σίγουρα εκατομμύρια. Σημειώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστια στρατιωτική παρουσία ε, από αυτά που βλέπουμε έτσι ποιος ξέρει τι γίνεται παραμέσα στην ενδοχώρα και μιλάμε ακριβώς για αυτήν την λεγόμενη συνοριοποίηση οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Την άλλη καλωσορίζουμε τα βήματα που κάνει η Γεωργιανή πλευρά για να βοηθήσει τον κλεισμό είτε μιλάμε για την Απχαζία είτε για την Νότια Σετία αν και στην Νότια Σετία δεν έχουν απομείνει τόσοι και όσοι έχουν απομείνει είναι στο πλευρό των ε, ρωσικών δυνάμεων Οπότε πρέπει νομίζω να καλωσορίσουμε κι εμείς οτιδήποτε συνεισφέρει στο να δείχνουν ότι ανήκουν στην Γεωργία είτε μιλάμε για ιατρικές υπηρεσίες είτε για οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα να βοηθηθούν μια συνεισφορά νομίζω πρέπει να τα δούμε θετικά. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει η δέκατη επέτειος χωρίς να κάνουμε μία δήλωση. Και όπως έγινε και τον Αύγουστο, θα πρέπει να προετοιμάσουμε κάτι στην Ολομέλεια του Ιουλίου γιατί η κατάσταση έχει παγώσει επί τόπου αλλά πρέπει να την θυμόμαστε και να αναφερθεί δημοσίως. Αυτό το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον, πέρα από το ότι οι δικοί μας περιγράφουν την κατάσταση, θα ήθελα να μάθω τι προτείνουν στους, ρο... στους με συγχωρείτε, τι πρέπει να κάνουν ή να μην κάνουν στο μέλλον και βεβαίως τι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για να προχωρήσει η κατάσταση και κάποια στιγμή όταν η Ρωσία θεωρεί ότι της κοστίζει πολύ τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε αυτή την διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον συνάδελφο, τον κύριο Περίμ, τον οποίο ούτως ή άλλως θα συναντήσω και απόψε και αύριο στην, ε, κοινοβουλευτική, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Σύνδεσης και στηρίζουμε και εμείς ε, την ιδέα ενός ψηφίσματος ε, του Κοινοβουλίου τον επόμενο μήνα. Η γεωργία, όπως υπόθηκε, κάνει πολύ καλή δουλειά, διατηρεί τις ανθρώπινες επαφές. Η νευτική πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει ε, μέσω του Κοινοβουλίου και νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, να δούμε πώς θα το στηρίξουμε, γιατί είναι αξιοθαύμαστο το ότι η κυβέρνηση ε, επιδεικνύει τέτοια βούληση για στενές ε, σχέσεις σε μια κατάσταση οπωσδήποτε πολύ δύσκολη προφανώς. Επίσης, όπως είπε η Πρόεδρος, ε, η Επιτροπή μας θα επισκεφτεί την Γεωργία την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου και θα μας βοηθούσε και πάλι να ακούσουμε κάποια σχόλια από εσάς όσον αφορά το πώς θα μπορέσουμε ακριβώ να έχουμε μια επίσκεψη με τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Κάποιες ε, συστάσεις δηλαδή για να έχει κάποιο όφελος αυτή η επίσκεψη. Το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας αναφέρθηκε επίσης Τι στήριξη λοιπόν θα μπορούσαμε να δώσουμε για την συνεργασία με την Ρωσία και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε η Λόρενς Μερντιστ για την ευελιξία γιατί βεβαίως είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα ώστε η αντίδραση πρέπει να είναι και αυτή η περίπλοκη. Προφανώς έχουμε τις συζητήσεις που θα γίνουν εδώ για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ήθελα και να μου απαντήσετε, αλλά και να σκεφτείτε μακροπρόθεσμα τι θα πρέπει να δούμε στο πλαίσιο αυτής της γραμμής του προπολογισμού στο μέλλον, αναγνωρίζοντας αυτό το οποίο είπατε για την ευελιξία. Και τέλος, να λάβω αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος, μια που είστε εδώ θα ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση για την παρέτηση του Πρωθυπουργού της Αρμενίας και για το τι συμβαίνει και στην Αρμενία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Στέτινα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω την γλώσσα μου, βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Η συζήτησή μας έχει τίτλο «Κατάσταση ασφαλείας στον Νότιο Κάφκασο» και συγκεκριμένα στην Γεωργία. Το αντιλαμβάνομαι ότι ε, είναι η δέκατη επέτειος της κατοχής της Νότιας Οσετίας τον Αύγουστο. Γι' αυτό εστιάζουμε ιδιαιτέρως στην Γεωργία. Θα ήθελα όμως, όπως ε, και η συνάδελφος, να πω ότι πρέπει σήμερα, και θα ήθελα μία απάντηση, από τους ειδικού να μάθω εάν ο Πρωθυπουργό Σαρκισιάν ε, και η παρέτησή του ε, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση ασφαλείας σε ολόκληρο τον Νότιο Κάφκασο, όπως επιδεινωθούν δηλαδή οι σχέσεις ε, με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ κύριε Κόμες. Ευχαριστώ για τη διοργάνωση της συζητήσεως Υποστηρίζω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για τη δήλωση που κάνει το Κοινοβούλιο επί τη ευκαιρία της δεκάτης επαιτίου. Και πράγματι, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της Γεωργίας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Γεωργία να μας πλησιάσει. Ήμουν επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας μας στις τελευταίες εκλογές και παρακολουθούσα τη δημοκρατική πρόοδο, τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος, τη λογοδοσία και εκεί μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά και το χρήμα μπορεί να βοηθήσει διότι βέβαια σχετίζεται πολύ με τις νέες πρακτικές, νέο διάλογο, διάδραση με τους διάφορους φορείς, τον ελεγκτικό ρόλο του Κοινοβουλίου, λειτουργία του δικαστικού κλάδου κλπ. Κατανοώ τα αναφερθέντα από τον κύριο Πχότσκης περί δράσεων των Ρώσων που κινούνται ως κατσαπλιάδες που έχουν σαν στόχο στρατηγικό δάση να προβάλλουν αυτή την ισχύ και πέρα από τη Γεωργία. Γι' αυτό είναι σημαντική η Γεωργία και πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά που κάνει ο πληθυσμός της Γεωργίας για να απορρίψει τους Ρώσους κατσαπλιάδες και την επιθετικότητά τους και την κατοχή των εδαφών τους. Ο Μάικλ Γκάλερ αναφέρθηκε στη σημασία της ιατρικής περίθαλψης των ανθρώπων που έρχονται από την Απκασία. Είδα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα στην Κύπρο. Η Νότια Κύπρος προσφέρει ελεύθερη διδασκαλία στους ανθρώπους από τα βόρεια κατεχόμενα εδάφη. Και κατόρθωσε έτσι να έχει μια ενδιαφέρουσα ροή ανθρώπων που έρχονται από τα βόρεια κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου και πάνε στην Ελεύθερη Κύπρου. Έχει στρατηγική σημασία η ρωσική γλώσσα. Αυτό, αυτός είναι ένας παράγος που υπόψη. Σε αυτό το πλαίσιο, τι ρόλο παίζει η Εκκλησία γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ θετικός. Και οι κοσμικές αρχές δεν αντιδρούν επαρκώς. Και κάτι άλλο. Εγώ συμπαραστέκομαι στο λαό της Γεωργίας. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν, όπως η δολοφονία και τα βασανιστήρια του κυρίου Τατνασβίλη, η Ρωσία αυτοπυροβολείται στο πόδι. Διότι έτσι οι Γεωργιανοί στρέφονται κατά αυτών των δράσεων των Ρωσικών. Υπάρχουν κάποια συμφέροντα ΜΚΟ, επιχειρηματικά συμφέροντα και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν συμφέροντα που εθελοτυφλούν όσον αφορά αυτά τα επεισόδια. Αυτό δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Δεν αφορά μόνο το να σταματήσουμε τη Ρωσία που φέρεται ως κατσαπλιάς επιτιθέμενη και προβάλλοντας ισχύ. Επίσης, πρέπει να απαλλαγούμε από τη ρωσική αντιμετώπιση των προβλημάτων εντός της Γεωργίας. Και σχετικά με αυτό δεν μπορώ να σιωπήσω. Είχαμε άλλη υπόθεση που καλύφθηκε από ψήφισμά μας. Απαγωγή του κυρίου Αφγάν Μουκαλή, ε, δημοσιογράφου του Αφγανιστάν, που τότε Λοιπόν, εγώ ταράχτηκα, διότι εντωμεταξύ η συνέντευξη του κυρίου Αφκάν Μουκτάλη λέει ότι υπήρξε ε, συνεργασία, υπήρξε συνενοχή με τους Ρώσους. Και ο Πρωθυπουργό συνεργάστηκε και ο πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Ιβανισβίλης συνεργάστηκε. Αυτό απαιτεί, αυτή η ε, υπόθεση απαιτεί κοινοβουλευτική έρευνα στη Γεωργία και υποστηρίζουμε το Κοινοβούλιο της Γεωργίας σε αυτή την έρευνα. Δεν αρκεί να απαλλαγούμε από τη Ρωσία πρέπει να απαλλαγούμε και από τη ρωσική νοτροπία και τον τρόπο δράσης κατά την άποψή μου. Αυτό διακυβεύεται όταν μιλάμε για, το, για την προσέγγιση της Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ακολουθήσει δημοκρατικό δρόμο. Αυτά θα ήθελα να ακούσω και τους εμπειρογνώμονές μας για την Αρμενία, τι έχουν να μας πούν, και για το Αζερμπαϊτζάν. Διότι βεβαίως δεν μπορούμε να παραμελήσουμε το ότι Πολύ σοβαρές αποκαλύψεις έγιναν ε, αρχές εβδομάδας στην έκθεση που διαβάσαμε, όπου οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν ένεργα προωθούσαν τη διαφθορά και των μελών του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαίων και των αξιωματούχων για να καλύψουν τη χειραγώγηση που άσκησαν σοφά τις εκλογές. Και σοβαρότατες αποκαλύψεις από τις δικές μας έρευνες για τη Μάλτα και το κράτος δικαίου στη Μάλτα και πώς εμπλέκεται το Αζερβαϊτάν στο ξέπλυμα χρήματος που αφορά το σκάνδαλο στη Μάλτα και σχετίζεται με τη δολοφονία Ευρωπαίας δημοσιογράφου ε, στην, της κυρία Γκαλίσια στην Μάλτα. Okay. It was the... Ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία παρέμβαση από Ευρωβουλευτή για αυτή τη συζήτηση. Και τώρα, οι ομιλητές μας θα απαντήσουν τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε το διευθυντή, τον κύριο Μέρεντιφ. Ο κάθε ένας από τους ομιλητές έχει έξι λεπτά για να απαντήσει. Ο κύριος Μέρεντιφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας για τα πολύ σωστά σχόλια και ερωτήσεις. Ε, πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσω τον κατηγισμό ερωτήσεις σε έξι λεπτά. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που είναι στα αριστερά μου και θα απαντήσει στα πιο πολιτικά ερωτήματα που θα καλύψω στα εξι λεπτά που έχω, ειδικά για τα θέματα της Αρμενίας πιο λογικό να σε απαντήσει η υπηρεσία εξωτερική δράση. Ούτω ή άλλω συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Ο λόγο που εστιάζουμε στη Γεωργία ε, είναι ότι δεδομένου του τίτλου ε, ήταν πολύ φιλόδοξο το σχέδιο να καλύψουμε όλε τι χώρε. Για την Αγκόρνο Καραμπάχ θα χρειαζόμασταν ε, μία χωριστή συνεδρίαση. Ένα βασικό θέμα ήταν ποιος είναι ο πιο χρήσιμος τρόπος για να δράσουμε, όχι μόνο μέσω μιας αποστολής. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, ειδικά για τη Γεωργία, αναφέρατε τις, ρωσικές, τις γεωργιανές αρχές, όλοι όσοι βοηθούν να προωθηθεί μια κουλτούρα και μια νοοτροπία ε, επικοδομητικού διαλόγου, που δεν αποκλεί κανένα, συνειδητοποιούν ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα αυτό. Όλοι ξέρουμε από ίδια πείρα σε διάφορες συγκρούσεις ότι πάντα υπάρχει κάποιος που έχει πιο σκληρή ρητορική και που επηρεάζει τον πληθυσμό και τα μυαλά του κόσμου και δημιουργεί διάθεση για αλλαγή ε, μάλλον και το να επηρεάσει τα μυαλά του κόσμου και να το δημιουργήσει διάθεση για αλλαγή, είναι σημαντικό να το κάνει μέσω διαλόγου. Η οικονομική υποστήριξη φυσικά ε, θα επηρεαστεί από τις δυναμικές που υπάρχουν στη χώρα. Ε, η αποστολή μας, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης κτλ. Τα λαμβάνουν όλα αυτά τα, πράγματα υπόψη και προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για επαφή. Ε, μιλήσαμε πολύ λοιπόν για θέματα ασφάλειας, ε, κυρίως για θέματα στρατιωτικής φύσης ασφάλεια. Ε, αλλά κάποιοι αναφέρθηκαν και στις ε, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο. Και πρέπει να υπάρχει διάθεση λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με όλου του πολίτε τη Γεωργίας. Εμεί από πλευράς Ευρωπαϊκή Ανώσης έχουμε μια διαρκή διαδικασία να ενημερωνόμαστε και να είναι όσο το πιο επίκαιρη η παρέμβασή μας. Και γι' αυτό ακριβώς σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την προσκλησία σας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να αντιδράσουμε ιδέες ε, για μια κατάσταση που μπορεί να αλλάζει πολύ γοργά. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο παγωμένος, ε, παγωμένη σύγκρουση, γιατί νομίζω ότι δεν καλύπτει καμία από τις ε, συγκρούσεις της περιοχής. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς η τα πρόσφατα γεγονότα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν την σύγκρουση αυτή παγωμένη. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη γλώσσα της Συνόδου Κορυφής που είναι ανεπίλητη. Τώρα, όποιο και αν είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε αυτό είτε το επόμενο, όποιο και αν είναι, και για να προσέξω λιγάκι πώς θα το θέσω εδώ, θα σας έλεγα ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίσης χρειάζεστε δυνατότητα γρήγορης απόκρισης, έγκαιρης απόκρισης και κάποια ευελιξία σε ό,τι αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης παρέμβασή σου. Καταλαβαίνω ότι για τις δημοσιονομικές αρχές αυτό είναι μια πρόκληση. Αλλά είναι σημαντικό για να είναι ε, επιτυχής η διαμεσολάβηση εγώ, ας πούμε, ε, συμμετείχα ε, στο διάλογο ε, Πριστίνας Βελιγραδίου όταν δημιουργήθηκε. Δεν υπήρχε αυτή η κατανόηση από πολλές πλευρές. Ε, αν υπήρχε μια διάθεση προς μια τέτοια κατεύθυνση, θα ήμασταν πολύ πιο ε, επιτυχείς. Νομίζουμε ότι διδασκόμαστε από κάθε σύγκρουση. Βεβαίως κάθε σύγκρουση είναι διαφορετική. Αλλά παρόλα αυτά κάποια πράγματα προσπαθούμε να τα μάθουμε και να τα εφαρμόσουμε στην επόμενη φορά. Αυτό που κατάφερα εγώ στη Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ με το εργαλείο Ευρωπαϊκής Γειτονίας είναι ότι σε οποιοδήποτε τομέα και αν μιλάμε η συμμετοχή μας επί μακρόν, ας πούμε, ε, σε μια διαρκή σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Παραδείγματος χάρη εδώ με τη γεωργιανή κυβέρνηση για θέματα ε, ασφάλειας. Έχουμε ένα διάλογο που δεν είναι μεμονωμένος, ε, σε μια παρατεταμένη σύγκρουση θα πρέπει να παρεμβαίνεις σε πολλά πράγματα. Όχι μόνο στην ασφάλεια. Ε, γεωργία, υγεία, ε, εκπαίδευση. Το σημερινό εργαλείο που συνεισφέρει στην σταθερότητα και την ειρήνη είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μαθαίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Εγώ αυτά έχω να πω. Και ένα τελευταίο, πραγματικά τελευταίο σημείο για την κυβερνοασφάλεια. Πολύ σημαντικό θέμα, μεγάλη προϋπόθεση και θα είναι και θέμα του πακέτου που σας παρουσίασα, που ετοιμάζεται, και η στρατηγική επικοινωνία με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Γεωργίας. Κάτι που θα συνεχιστεί και αυτό είναι προϋπόθεση. Υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσα να πω, αλλά δεν έχω χρόνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόρενς. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές για τις ερωτήσεις σας και ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω μέσα σε έξι λεπτά. Θα ξεκινήσω από την Αρμενία γιατί δεν έχει απαντηθεί. Ε, εγώ ήμουν στην Αρμενία μέχρι πέρσι τον Σεπτέμβριο. Πέρασα τέσσερα χρόνια εκεί και κάθε χρόνο ε, έβλεπα κάποιες διαδηλώσεις αλλά φέτος είδαμε ένα νέο επίπεδο αν θέλετε στις ε, διαμαρτυρίες είχαμε το ενδιάμεσο αποτέλεσμα που οδήγησε στην παρέτηση του νέου πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου. Σημειώσαμε την ε, παρέτηση αυτή του κυρίου Σαρκισιάν. Κατά την άποψή μας έχει μεγάλη σημασία να ολοκληρωθεί και να επιληθεί σύντομα η κατάσταση και να ολοκληρωθεί ο εθνικός διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεχίσει την συνεργασία της με την Αρμενία να εφαρμοστεί η φιλοδοξία ατζέντα που έχουμε σύμφωνα με την ενισχυμένη Συμφωνία Συνεργασίας που ενέκρινε ομόφωνα το Κοινοβούλιο της χώρας το 2018 και ελπίζουμε να εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εδραιωθεί η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δημιουργηθεί έτσι ένα σύστημα ε, οικονομικής ευημερίας. Τώρα, για ένα ερώτημα το οποίο συζητήθηκε νομίζω εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αρμενία, το οποίο αφορά την Ρωσία και τον αντίκτυπο της λεγόμενης βελούδινης επανάστασης στις σχέση με την Ρωσία και νομίζω πως ε, αυτό το οποίο είπε ο επικεφαλής των διαδηλωτών χτες ε, στην συνέντευξη τύπου είναι κάτι το οποίο απαντά είπε ότι δεν είμαι υπέρ της Ρωσίας ή υπέρ της Δύσης είμαι υπέρ της Αρμενίας και ε, πράγματι βλέπουμε ότι οι διαμαρτυρίες αυτές σχετίζονται με μια καθυστερημένη αντίδραση που υπήρχε μετά τις εκλογές ε, το ότι ο πρόεδρος κατέλαβε την θέση του Πρωθυπουργού ε, κατά το οποίο προφανώς δεν άρεσε σε πολλούς και πολλούς νεαρούς που βγήκαν στους δρόμους επίσης ε, το θέμα είναι και ζήτημα οικονομικής ευημερίας ε, του μέλλοντος που βλέπει ο κόσμος ή δεν βλέπει στη χώρα ή μεταρρυθμίσεις ε, και στον τομέα της του καταπολέμησης της διαφθοράς και των κατσαπλιάδων. Δεν πρέπει λοιπόν να μεγενθύνουμε τα πράγματα πέρα από την σωστή τους διάσταση ότι υπήρχαμε και στο παρελθόν ανάλογες διαμαρτυρίες σε άλλες χώρες. Τώρα για τον Αγκόρνο Καραμπάχ βεβαίω υπάρχουν αναφορές ε, των ΜΜΕ για κινήσεις ε, στρατευμάτων, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί νομίζω. μη βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και βεβαίως ε, καλούνται, βλέπουμε εδώ πέρα όλες οι πλευρές να μειώσουν τις εντάσεις και αναμένεται μια συνάντηση των μερών των στομότερο δυνατών για να ενταθούν οι διαπραγματεύσεις για να βρεθεί μια μόνιμη λύση στην σύγκριση. και όπως ξέρετε η θέση μας είναι ότι υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των συμπροέδρων της ομάδας του Μίνσκ. Επίσης, όπως ανέφερε και η συμπρόεδρος ε, της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ότι το status κουβό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήταν κάτι το οποίο διαβίβασε και ο πρόεδρος Τούσκ ε, ε, στους πρόεδρους Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν όταν ήρθαν στις Βρυξέλλες και τα επανέλαβε και η κυρία Μογκερίνη. Επίσης, είδαμε και κάποια δυναμική στις διαπραγματεύσεις του μηχανισμού της ε, Κρακοβίας και αν μου επιτρέπετε τώρα θα στραφώ στην ε, Γεωργία. Δύο ερωτήσεις έγιναν. Τι μπορεί να κάνει παραπάνω η Γεωργία, τι μπορεί να κάνει παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμά μας στη Γεωργία ήταν πάντα ότι υπάρχουν δύο επίπεδα στην σύγκρουση, ένα με την Ρωσία και ένα με την διεθνή κοινότητα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γι' αυτό ακριβώς καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία για την ειρήνη και ενθαρρύνουμε τη Γεωργία να συνεχίσει αυτήν την ε, πορεία παρά το ότι έχουν πει ήδη ότι δεν ενδιαφέρονται αλλά μια τέτοια διαδικασία βέβαια απαιτεί χρόνο και πολιτική βούληση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουμε με την πολιτική μη αναγνώρισης και νομίζω ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει εδώ πέρα να δούμε ακριβώ ε, τις ε, δυνατότητες μιας ε, συμφωνίας ελευθερού για την περίπτωση Τζίλιεφ επίσης το παρακολουθούμε στενά όσον αφορά τον Μουχτάλη ε, έχουμε ακριβώς ε, και την απάντηση που έδωσα εντός του Κοινοβουλίου πρόσφατα για τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σας διαβεβαιώ ε, πως είμαστε σε επαφή και με τις αρχές του Αζερβαϊτζάν. Να έρθω λοιπόν στο Αζερβαϊτζάν, ένα τελευταίο σημείο για το πλυντήριο το λεγόμενο σημειώσαμε την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης γιατί είδαμε ότι ε, λέει εκεί πέρα η έκθεση ότι παραβιάστηκαν κάποιοι κανόνες δεοντολογίας η έκθεση έρχεται μετά από μια αξιόπιστη και ενδελεχή έρευνα και ζητάει από το Κοινοβουλίο να αντιδράσει σε αυτές τις κατηγορίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την εφαρμογή από το Συμβούλιο της Ευρώπης των συστάσεων αυτών που περιέχει έκθεση. Αυτό θα είναι σημαντικό για την σταθερότητα και αξιοπιστία της κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μάντα Πολ. Να σχολιάσω σύντομα το θέμα της Αρμενίας πολύ θετικά τα τεκτενόμενα στην Αρμενία. Συγχαρητήρια όσον αφορά την αρμενική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών στην Αρμενία, έγινε ισχυρός παράγων για την αλλαγή με έναν τρόπο ανέφικτο προηγουμένω. Διαδήλωσαν, έδειξαν ότι δεν δέχονται αυτού του είδους την κυβέρνηση που επί δεκαετίες επικρατούσε στην Αρμενία, ότι επιθυμούσαν δημοκρατική χώρα, κράτος δικαίου και αυτό είναι πραγματικά θετικό αλλά πόρα απέχουμε από το τέλος του παιχνιδιού διότι ακόμα διεξάγονται διαμαρτυρίες στους δρόμους και δεν είναι το τι πρόκειται να συμβεί. Ελπίζω ότι οι αρμενικές αρχές θα συνεχίσουν να μην χρησιμοποιούν δύναμη σαν κατσαπλιάδες γιατί είναι σημαντικό να το κάνουν αυτό. Διότι όταν χρησιμοποιείται δύναμη στην επόμενη φάση θα έχει σοβαρές συνέπειες. Όσον αφορά τη Ρωσία, οι Ρώσοι ήταν αρκετά σιωπηλοί, διότι η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχουν αναμειχθεί. Έχει φύγει ο Πρωθυπουργό, αλλά δεν ήταν ο μόνο ε, παράγων στο αρμενικό πολιτικό προσκήνιο που εκπροσωπεί ρωσικά συμφέροντα. Η Ρωσία παίζει προσεκτικά ε, στο παρασκήνιο το παιχνίδι, διότι οι Ρώσοι δεν θέλουν να δημιουργήσουν αντιρωσικά συναισθήματα έντονα στην Αρμενία, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, όπου θεωρούνται οι Ρώσοι σαν κατσαπλιάδες της περιοχής. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και θα είναι πολύ σημαντικό και κατά κάποιο τρόπο θα αυτό θα επηρεάσει και τον Αγκόρνο Καραμπάχο. Ο πρόεδρος Αλίευ θα έχει άλλο διαπραγματευτικό εταίρο στην ειρευτική διαδικασία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και ελπίζω να μην υπάρξουν ανόητες εξελίξεις, να μην προσπαθήσει κανείς να ωφεληθεί με άλλα λόγια από το δημιουργηθέν κενό ε, που περιστρέφεται γύρω από τη σύγκρουση που είδαμε κατά παρελθόν. Ελπίζουμε λοιπόν να μην υπάρξουν σοβαρές παραβιάσεις της καταπαύσεως του πυρός. Όσον αφορά τι παραπάνω μπορεί να κάνει η Γεωργία. Νομίζω ότι η Γεωργία θα πρέπει να βασιστεί επί των ίδιων επιτευχθέντων και να συνεχίσει να είναι δραστήρια και δημιουργική όσον αφορά το πλησίασμα στον πληθυσμό της Νότιας Οσετίας και της Απκαζίας. Τι ούτω τρόπος να κινηθεί με τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων στη Γεωργία χρειάζεται ένα ενιαίο μέτωπο, ε, πολυσχηδές, και η κοινωνία των, της Γεωργίας να γνωρίζει ακριβώς τι προσέγγιση ακολουθείται, να μην υπάρχει περιθώριο παρερμηνιών και παρεξηγήσεων που μπορεί να αποτελούν πρόβλημα. Και να επαναλάβω αυτό που είπατε για την Κύπρο. Πιστεύω ότι η Κύπρος είναι ένα καλό μοντέλο, όχι για επίλυση των συγκρούσεων, δεν τα καταφέραμε ακόμα εκεί, δεν φτάσαμε εκεί, αλλά πλευράς εμπειριών και βελτίστων πρακτικών μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτά που πέτυχαν οι δύο κοινότητες. Ίσως να μην έχουν μια λύση, αλλά τα πάνε καλά μεταξύ τους. Χιλιάδες Κύπροι πάνε από τη μια πλευρά στην άλλη, ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση, αλλά μπορούμε να αντλήσουμε κάποια μαθήματα από εκεί. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίζει παντιοτρόπως την πρωτοβουλία, τις πρωτοβουλίες της Γεωργίου. Αλλά μετά τη δέκατη επέτειο του πολέμου κάτι πρέπει να υποθεί και ίσως κάποιος προβληματισμός επί περαιτέρω ενεργειών για να σταματήσουν οι μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεχιζόμενη συσσόρευση στρατευμάτων. Ξέρω ότι δεν είναι καλό αυτό που λέω, αλλά πιστεύω ότι το θέμα των κυρώσεων των κυρώσεων πρέπει να τεθεί επιτάπητος, διότι δεν καταλαβαίνω διότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε μια σύγκρουση στην Αρμενία και σε παρόμοια περιπτώσεις και δραστηριότητε όσον αφορά ε, την παραβίαση της κυριαρχία της γεωργία. αυτό δεν τίθεται σαν θέμα. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου δημοφιλές να συζητά κανείς για κυρώσει, αλλά θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ο κ. Πορκίτζα, λόγο. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω με τις διαδηλώσει και να πάμε μετά Ρωσία-Αρμενία, τι σχέσει Μπακού και μετά θα ολοκληρώσω με τα σχόλια περί Γεωργίας. Αρχικά Συμφωνώ με τους άλλους. Ό,τι συνέβη στην Αρμενία είναι σημαντικότατο, όχι μόνο την Αρμενία, αλλά για όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Μερικά σχόλια έχω όσον αφορά την φύση των διαμαρτυριών και των δηλώσεων. Βασικά, ακόμα και εντός της Αρμενίας είχε τον τίτλο σαν διαμαρτυρία της νεολαίας. Υπάρχει ένα στοιχείο γενιάς μέσα σε αυτό και να το προσέξουμε. Άλλο, κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι για τις διαμαρτυρίες και η αίσθηση ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Βλέποντας τι λένε οι εμπειρογνώμονες, διαβάζοντας τα άρθρα, υπάρχει το κοινωνικονομικό στοιχείο. Η Αρμανία συνήψε τη συμφωνία για το εμπόριο, ενστερνίστηκε το ευρωπαϊκό μονοπάτι. Με περιορισμένο, πολύ περιορισμένο τρόπο. Λόγω της Ευρασιατικής Οικονομικής Ενώσεως δεν καταφέραν να ξεγελάσουν τον πληθυσμό. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Άρα έχει νόημα τελικά να επενδύει κανείς στη χώρα μεγάλο σφάλμα του Σαρκισιάν. Διότι υπερέβαλε στο παιχνίδι που έπαιξε. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να εξετάσουμε κάποια στοιχεία. Αφορά αλλαγή, πραγματική αλλαγή της εξουσίας είναι διακοσμητικού χαρακτήρα η αλλαγή. Θα δούμε αν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Το θέμα είναι ποιος θα χειρίζεται τις εκλογές. Όλοι συμβιβάστηκαν ότι πρέπει να ξαναποφανθεί ο λαός. Υπάρχουν ε, διαμάχες για το θέμα. Ποιος θα διαξάγει τις εκλογές, η κυβέρνηση, η υπηρεσιακή κυβέρνηση, όπως θα την αποκαλέσουν, προσωρινή κυβέρνηση, τις οποίες θα ηγούνται οι επικεφαλής των ε, διαδηλώσεων. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είναι λογικό να μην μειωθούν οι αριθμοί που διαδηλώνουν, εκείνοι που διαδηλώνουν. Να μην θεωρηθεί ότι ε, έχουν πετύχει κάτι, υπάρχει κάτι κεκτημένο, κάποιο κεκτημένο. Ακούγονται θριαμβολογίες και δεν πρέπει να ακούγονται τώρα ακόμα. Ρωσία-Αρμενία. Πώς αυτή η σχέση επηρεάζει τις εξελίξεις. Κάποια σημαντικά σημεία να θυμόμαστε. Η ερμηνεία θεωρείται απεκλεισ... εγκλωβισμένη μάλλον. Και ίσως η αδίποτε αλλαγή δεν μπορεί να μεταφραστεί σε επαναπροσανατολισμό της θέσης της ή τουλάχιστον ξαφνική αλλαγή, ίσως να χρειαστεί χρόνος. Γιατί είναι θέμα οικονομίας και εμπορίου που εξαρτάται πολύ από τη Ρωσία, ενεργειακά εξαρτάται κατά πολύ από τη Ρωσία, κυρίως για το φυσικό αέριο, αφορά το Καραμπάχ, την επικράτεια της Γεωργίας. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Σίγουρα πρέπει να τα εξετάσουμε. Θα χρειαστεί χρόνος. Για τις διαμαρτυρίες, η ρωσική σιωπή, όσον αφορά τις διαδηλώσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα η σιωπή. Άλλοι θεωρούν ότι είχαν φυσικάσει, δεν έβλεπαν θα συμβεί κάτι. Άλλοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή. Αληθεύουν και τα δύο. Υπάρχουν στοιχεία και από τι δύο πλευρέ. Υπάρχουν πάντα μαθήματα που μπορεί να μάθει κανεί, ιδιαίτερα εδώ. Για τη Γεωργία, τι μπορεί να γίνει και από τι δύο πλευρέ. Συμφωνώ με την αξιολόγηση που εκφράστηκε. Δεν αφορά μόνο καταπολέμηση της ε, Ρωσίας διεθνώς, αλλά και εντός Γεωργίας. Τι μπορεί να γίνει. Πρωτίστως, θέμα κόστους για τη Ρωσία, να κοστίζει περισσότερο στη Ρωσία. Ε, συνεχούς προσπάθειας, συνέπειας, σαφήνεια πολιτικής διπλωματικής γλώσσας και δράσεως. Οι κυρώσεις είναι σημαντικότατες. Η, η Γεωργιανή κυβέρνηση γιατί δεν πιέζει για κυρώσεις σε συνάρτηση με τις κατεχόμενες περιοχές. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν ακούω πολλέ φωνές πάνω σε αυτό την τυφλίδα. Θα πρέπει να συνδεθούν με το θέμα και κυρώσει. Δεν είναι δημοφιλές θέμα κυρώσει, το ξέρω. Αλλά είναι σημαντικότατο ζήτημα. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Το UMM πρέπει να συνεχιστεί επιτόπου. Θα γίνουν ακροάσεις. Να συνεχιστεί η υποστήριξη της Γεωργίας. Αυτή η δήλωση τη Ρωσία για τιμή χρήση ισχύω και δύναμη δεν πρέπει να Διότι η Γεωργία έκανε μονόπλευρη δήλωση και δέσμευση, δεν έκανε κάτι παρόμοιο η Ρωσία. Η αδίποτε αλλαγή που σχετίζεται με τη Γενέβη, όπως προβλήθη εσφαλμένα, δεν θα έχει νόημα χωρίς σαφή δέσμευση της Ρωσίας για τιμή χρήση βίας. Τι μπορεί να κάνει η Γεωργία. Πολλά μπορεί να κάνει. Ανέφερα κάποια στοιχεία. Έχει κι άλλο πρόβλημα. Δεν πολεμά τη Ρωσία αρκετά στο εσωτερικό της. Να αναφερθώ στο πώς βλέπει η Γεωργία την ανάπτυξή της και την εξέλιξή της. Πολλοί στην Τυφλίδα θεωρούν ότι η Γεωργία είναι πρώτη όσον αφορά τις επιδόσεις της και αρκεί. Υπάρχει μια σχετικιστική προσέγγιση και δημιουργούνται προβλήματα. Μιλάμε για πρόβλημα πλουραλισμού. Η Γεωργία δεν έχει ισότιμους όρους πολιτικά. Υπάρχει μεροληψία υπέρ του κόμματος που είναι στην εξουσία. Έχουμε ένα στοιχείο, πολιτικό στοιχείο, κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, αδύναμη ηγεσία, άτυπη διακυβέρνηση, τεράστιο πρόβλημα για τη Γεωργία, εξακολουθεί έλλειψη λογοδοσίας, μέσα ενημέρωσης και πλουραλισμός των ΜΜΕ, δικαστικός κλάδος, πέραν αυτών. Η Γεωργία και οι Γεωργιανοί αξίζουν προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πολλά τα προβλήματα θα σχετίζονται με προοπτικέ ε, προσχώρηση. Να αναγνωριστεί δεν σημαίνει να γίνει μέλο. Δεν αφορά μόνο τη Γεωργία. Εν γέννη. Δεν είναι δημοφιλέ θέμα, το ξέρω. Εν γέννη, μια προπτική τέτοια θα είναι διαφορετικό ποιοτικό επίπεδο ε, του δέλεαρ που μπορεί να, να προσελκύσει την ελίτ. Βλέπουν τη συμφωνία σύνδεσης σαν μια γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι έχουν τα πράγματα. Okay. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε παρά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, πανελίστες μας. Παρακαλώ χειροκροτήστε. Ευχαριστώ. Ε, μην φύγετε από την αίθουσα, έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη.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 αδελφοί, παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την κυβερνοασφαλεία των αποστολών ε, και επιχειρήσεων της ΚΟΠΟΑΑ και είναι χαρά μου να καλωσορίσω δύο διακεκριμένους ομιλητές και τον κύριο Στέφαν Χούμπερ, επικεφαλής ε, της ε, μονάδας στήριξης αποστολών ε, και τον κύριο Νιλπαϊρ που επίσης είναι επικεφαλής της μονάδας κυβερνάμινας. Κυβερνοάμυνα λοιπόν είναι το θέμα και θα ήθελα να δώσω λόγο μάλλον στην ομάδα πρώτα και μετά να ακούσω τις ε, σχετικές ε, ε, δράσεις που λαμβάνονται για να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας στις αποστολές. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα σας δώσω μια σύντομη εικόνα. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τις ε, υφιστάμενες αποστολές, έξι στρατιωτικές και δέκα πολιτικές. Οι πολιτικές αποστολές απασχολούν 2.000 άτομα, η μισή είναι αποσπασμένη από τα κράτη-μέλη, 500 είναι τοπικοί και οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι. Εν ολίγης, στις 10 αυτές αποστολές έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε πολύ λίγο κόσμο στα κεντρικά. Ιστορικά δηλαδή δεν είχε υπάρξει σε κεντρικό επίπεδο ικανότητα κληροφορικής. Αυτό έχει θετικά και αρνητικά στην περίπτωση ε, των πιθανών υποθέσεων, επιθέσεων η αποκέντρωση είναι οπωσδήποτε ένα πλέον έκτημα έχουμε λοιπόν χωριστά δίκτυα που στείνει κάθε αποστολή χωριστά αυτό σημαίνει βεβαίω τους ε, υπάρχει διαφορετικός βαθμός προετοιμασίας και προσπαθούμε σταδιακά να τα φέρουμε όλα σε ένα υψηλό επίπεδο έχουμε όπως είπαμε δεδομένης της δομής ε, του συστήματός μας έχουμε μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε κάθε αποστολή κάθε αποστολή έχει τη δική της νομική προσωπικότητα Υπάρχουν λοιπόν συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με την ομάδα υπολογιστών ε, και υπάρχουν κάποια σημεία επαφής όπως έχουμε κάνει στην ΚΑΠΑΠΙΑΛΦΑΛΦΑ Έχουμε λοιπόν αφιερώσει μια θέση διοικητικού προσωπικού, ο ειδικό μας είναι εδώ στην αίθουσα και από όταν ήρθε αυτός ο ειδικό εναρμονίζουμε και ενισχύουμε τις αμυντικές δυνατότητες. Να προχωρήσω παρακάτω. Εργαζόμαστε επί τη βάση ενός εγγράφου που προετοίμασε η υπηρεσία και ενέκρινε η Πολιτική Επιτροπή και συμπληρώνει βασικά το προηγούμενο έγγραφο που είχε εγκριθεί αναφέρει συγκεκριμένα επιχειρησιακά βήματα υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει στρατιωτική και πολιτική συνεργασία και να αναγνωριστεί το ότι υπάρχουν διαφορετικά προφίλ κινδύνου και επιμελητίας γιατί έχουμε διαφορετικές πηγές ε, προϋπολογισμού και διαφορετικούς κανόνες επίσης. Σαφώς το έγγραφο αυτό έχει στόχο να είναι σε θέση επικεφαλής των αποστολών να δουν ακριβώς ε, τα ευπαθή σημεία σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες επιθέσεις ε, δηλαδή να υπάρξει μια αξιολόγηση κινδύνου και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθούν οι κίνδυνοι και βεβαίως ε, να ανακάμψουμε και από κυβερνοεπιθέσεις. Το έγγραφο αυτό είναι ένα έγγραφο ιδεών μας δίνει μια γενική εικόνα για τον ρόλο των κυβερνοπληροφοριών. Δηλαδή, Έχουμε λοιπόν πολλούς ειδικού εδώ, εξετάζουμε τις κυβερνοαπειλές, ειδικά στην φάση της προετοιμασίας νέων αποστολών, όσον αφορά την διαδικασία σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής το σχέδιο και η δήλωση προϋπολογισμού πρέπει να περιλαμβάνουν μέσα και δραστηριότητες από την αρχή της αποστολής ε, η κυβερνοασφάλεια είναι τμήμα των επιχειρήσεων. Βεβαίως το έγγραφο αφιερώνει και αποδίδει κάποια σημασία στην φάση της επαφής στην οργάνωση των ευθυνών και των δικτύων εκπαίδευση κατάρτιση, ασκήσεις, ε, κυβέρνηση και ανάπτυξη ε, δυνατοτήτων. Να σας δώσω τώρα μια εικόνα για την φάση της εφαρμογής ε, στις πολιτικές αποστολές. Όπως είπα έχουμε έναν ειδικό και ένα από τα κύρια καθήκοντα είναι οι επαφές ε, με τους ειδικού και έχουμε διασφαλίσει τώρα ότι έχουμε ένα, μια σύμβαση πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια κάτι το πολύ σημαντικό Μειώνεται έτσι η γραφειοκρατία και επιτρέπεται έτσι να έχουμε ένα υπόδειγμα στις διαδικασίες ε, προμηθειών. Βεβαίω κάθε επιχειρησιακό σχέδιο έχει αναφορά στο έγγραφο που ανέφερα πριν, αλλά τώρα μιλάμε για μια παράγραφο η οποία θα είναι πιο συγκεκριμένη και όσον αφορά τις ε, απαιτήσει ε, αναφέρω απλά τρία σημεία. Έχουμε την αξιολόγηση κινδύνου, το να υπάρχει κάποιο σημείο επαφής σε κάθε αποστολή για την κυβέρνηση ασφάλεια. Επίσης αναφέραμε, όπως είπαμε, τις ε, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών. Έχουμε την ομάδα αντίδρασης ε, σε δύο επίπεδα ε, υπηρεσιών. Το ένα είναι η δωρεάν πρόσβαση και μετά έχουμε και τις υπηρεσίες επιπληρωμή. Μιλάμε δηλαδή για τεστ διείσδυσης, όπως λένε οι ειδικοί, αξιολόγηση ευπάθειας και διαχείριση συμβάντων. Αυτά υπάρχουν ήδη στην αποστολή της Ουκρανίας και της Γεωργίας και πρέπει να πω ότι όλα αυτά είναι πολύ πρόσφατα από το τέλος του 2016 και εφαρμογή κυρίως το 2017. Οι πολιτικές αποστολές ε, εκπροσωπούνται στην ε, Task Force ε, και στον μηχανισμό κύβερνο διοίκησης. Πολύ σημαντικά όλα αυτά λόγω της διαφοράς στην φύση των συστημάτων πληροφορικής Όλα αυτά λοιπόν έχουν κάπως παρόμοιες δομές και κοινέ πλατφόρμες. Οι αποστολές αυτές τις πολιτικές έχουν τα δικά τους τοπικά συστήματα. Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή στο στήσιμο μιας πλατφόρμας για τις πολιτικές αποστολές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εντός του μηχανισμού διοίκησης και τέλος οι δεξιότητες κυβερνοασφάλειας που υπάρχουν πλέον στην περιγραφή των καθηκόντων για τους αρμόδιους πληροφορικής ε, και ασφαλείας. Οπότε είναι πράγματα τα οποία ε, κάνουν, ε, κάνουν και το τοπικό προσωπικό. Πάω στην περίπτωση της Ουκρανίας τώρα. Η περίπτωση της Ουκρανίας λοιπόν Είχαμε διάφορες ε, κυβερνοεπιθέσεις μετά τα γεγονότα του Μαϊντάν και της Κρυμαίας. η αποστολή έχει ένα σχέδιο προστασίας ε, με κυβερνοελέγχους και ανάπτυξη διάφορων δυνατοτήτων. Από την οργάνωση της αποστολής ε, υπάρχει προετοιμασία για κυβερνοεπιθέσεις από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η αποστολή. Και υπάρχουν και σχέδια ε, ασκήσεων για αντιμετώπιση περιπτώσεων κυβερνοεπιθέσεων. για τη διακυβέρνηση. Μάλλον το κείμενο που έχω μπροστά μου διαφορετικό από τις διαφάνειες. Υπάρχει ο σχεδιασμός και η εφαρμογή. Και μόλις τελειώσει, φτάνουμε σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, εσωτερικά τα πράγματα ε, ομαλά, αλλά σε επιχειρησιακό επίπεδο οι δραστηριότητες, δηλαδή, ε, σε ό,τι αφορά τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην τομέα της ασφάλειας, για αυτούς παρέχουμε κατάρτιση, ειδικά για τις διοκτικές αρχές. 40.000 ε, χρήστες ε, εκπαιδεύονται και περνάνε από εξετάσεις. Ε, γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης ασφάλεια για τις διοικητικές αρχές. Ο, γίνεται ένας ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων και το 2017 η ΙΟΑΜ υποστήριξε τις ε, διοικητικές αρχές Ουκρανίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας κατάρτιση. Χρησιμοποίησε μια εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Ήταν μια πολύ γρήγορη παρουσίαση που την έκανα πολύ αργά. Ο κύριος Νίλ Πάουερ, ε, επικεφαλής της ομάδας για την κυβερνοασφάλεια, ε, από πλευράς της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Καλησπέρα. Είμαι επικεφαλής της ομάδας στην διεύθυνση CIS. Θα σας μιλήσω λίγα λεφτά για τη στρατιωτική πτυχή της ΠΑ Μία ομάδα για την κυβερνό άμυνα δημιουργήθηκε με βάση τις, τους πόρους που έχουμε ε, το 2012. Ένα άτομο στην αρχή είχαμε, ε, μετά δυόμιση άτομα και αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον που υπάρχει στον τομέα αυτό, την αύξηση των απειλών όμως επίσης και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό. Γνωρίζουμε ότι τα συστήματα μας είναι διασυνδεδεμένα και στον πολιτικό τομέα, αλλά το ίδιο ισχύει και για το στρατιωτικό τομέα. Αυτά τα συστήματα πληροφορικής μας δίνουν τη δυνατότητα να, κάνουμε όλες τις, να προωθούμε τις δράσεις της ΚΠΑ. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε το πλαίσιο και βλέπετε την διοικητική δομή που υπάρχει, γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην ε, πολιτική πλευρά και στρατιωτική πλευρά και στην στρατιωτική πλευρά μεταξύ των ε, αποστολών και των επιχειρήσεων. Στα επιχειρησιακά επίπεδο έχουμε πέντε ε, αρχηγεία στα κράτη-μέλη. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό αρχηγείο, συν την εγκατάσταση στο Βερολίνο, καθώς και ένα κέντρο στην EUMS. Οι τρεις επιχειρησιακές αποστολές που είναι εκτελεστικέ αποστολές που είναι εξελίξει σήμερα έχουν υποστήριξη από τα έθνη που, τις, που υποφελούνται από αυτές. Ε, προστασία των δικτύων, επιστοποίηση, ασφάλεια. Είναι πολύ πιο έντονο το πλαίσιο από ό,τι στις αποστολές. Έχουμε τη Σοφία, την Αταλάντα, στο κέρας Αφρικής, ε, το αρχηγείο του Ινωμένου ε, Βασιλείου και η Αλθία στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Μέχρι πέρυσι οι αποστολές γινούσαν ανεξάρτητα. Ε, αλλά το κέντρο ε, στρατιωτικού σχεδιασμού που βλέπετε στη διαφάνεια ε, είχε θετικές επιπτώσεις συντονίζοντας τις δραστηριότητες αυτές. Είμαστε υπό εξέλιξη και δεν έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις στην οργάνωση. Μία από τις θέσεις είναι θέση υπευθύνου για την κυβερνοάμυνα. Παρέχουμε και πραγματογνωμοσύνη στην οργάνωση αυτή. Καθώς αναπτύσσεται η οργάνωση αυτή, βλέπετε τη δυνατότητα να βρούμε λύσεις και δυνατότητες που μέχρι στιγμή είναι απομονωμένε στι διάφορε αποστολέ. Στην MPCC βλέπετε και τη CPCC ε, για την πολιτική πλευρά σας, για την οποία σας μίλησε ο συνάδελφος και υπάρχει μια σχέση, ε, ένα, ένας πυρήνας ε, υποστήριξης και συντονισμού είναι η οργάνωση, ε, αλλά θα δημιουργηθεί μια πραγματική ε, οργάνωση με περισσότερες δυνατότητες. Επίσης, βλέπετε το δικό μας ρόλο να δούμε τις πολιτικές πριν από την έγκριση μιας επιχείρησης ή μιας αποστολής, κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να δούμε ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία ούτω ώστε ο διοικητής της, του επιχειρησιακού κομματιού να λάβει τις ευθύνε του. Αναπτύξαμε και μία ε, έννοια για την κυβερνοάμυνα. Ε, αυτό έγινε και το 2016. Εγκρίθηκε από την ε, στρατιωτική αποστολή τον Αύριο του 2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το έγγραφο είχαμε το σκοπό να εξετάσουμε τις ευθύνες, αρχές, διαδικασίες, ούτως ώστε να δώσουμε ε, καθοδήγηση στην ομάδα σχεδιασμού, ε, στο διοικητή της επιχείρησης για το τι έπρεπε να κάνει, τι πρέπει να λάβει υπόψη του όταν προετοιμαζόταν για μια πιθανή επιχείρηση ή αποστολή. Επίσης, ε, κάποιες κατευθυντήρες γραμμές προς τα κατημέλη κατά την προετοιμασία των δυνατοτήτων τους που μπορεί να απαιτηθούν στο μέλλον για αυτές τις αποστολές. Υπάρχει το θέμα της ορολογίας, ασφάλεια και κυβερνοάμυνα. Ε, το χωρίζουμε έτσι απλουστευτικά. Στην, ε, ε, η ασφάλεια αφορά το πολιτικό τομέα, ενώ η άμυνα αφορά το στρατιωτικό τομέα. Ε, έτσι περιγράφουμε τα πράγματα στο concept. Ε, φυσικά δεν υπάρχει τυποποιημένη ορολογία και ξέρετε ανάλογα με το κράτος μέλος και το σε ποιον μιλάτε, ε, υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο για να το εξετάσουμε. Πολύ σύντομα. Για το, την έννοια της κυβερνοάμυνας, ε, δεξιά βλέπετε τη δομή, ένα κατάλογο με τις δυνατότητες, την, ε, το δόγμα, το προσωπικό, ηγεσία, δραστηριότητες, τι, τι καλύπτουμε εκεί και αριστερά βλέπετε τις αρχές. Ε, βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για μια επιχείρηση αποστολή. Δεν μπορείς να προσθέτεις δηλαδή δυνατότητες ατελεύτητα, θα πρέπει να τα καθορίσεις αυτά από την αρχή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ε, πριν ξεκινήσεις μια αποστολή ή μια επιχείρηση. Η αξιολόγηση, οι πληροφορίες, ε, αξιολόγηση απειλής που πας, ποιο το περιβάλλον, και αυτά που είπε ο συνάδελφο. είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να ξέρεις ε, τι τι αντιμετωπίσει για να μπορείς να το αντιμετωπίσει. Προετοιμασία λοιπόν, σχεδιασμός, αλλά πρέπει να μπορείς να αντιδράσει και να επανέλθεις μετά από αποστολή. Χρειάζεσαι ανώτερους αξιωματούς που καταλαβαίνουν το περιβάλλον. Μιλήσαμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πολιτικό και στο στρατιωτικό σκέλος και υπάρχουν και νομικές πτυχές. Χρειάζεσαι νομομαθείς, νομικούς, κάτι, κάποιοι που καταλαβαίνουν το περιβάλλον, που μπορεί να υποδείξουν τη σωστή πορεία δράσης. Τι, αυτή δεν υπάρχει, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι η χρηματοδότηση. Έχουμε το μηχανισμό Αθήνα, για να ζητήσουμε χρηματοδότηση για τις δραστηριότητε. Ε, βάζουμε, ας πούμε, πριν την αρχή της αποστολής ε, ένα ποσό αναφοράς και ο διοικητής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η κυβερνάμενα έχει ληφθεί υπόψη, ούτε ώστε να έχουμε τους σωστούς πόρους. Και δεν μιλάω μόνο για τεχνολογία, μιλάω και για όλες τις υπόλοιπε πτυχές που αναφέρονται στα δεξιά, στην δεξιά στήλη. Πολύ σύντομα θα καλύψω τις ε, σημαντικές ε, επακόλουθες δραστηριότητε που προωθούμε και προωθήσαμε και προωθούμε εδώ και 15-16 μήνες. Ε, υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία ε, λειτουργίας, ε, συνεργασία με το OHQ και το MPCC. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λογοδοτούμε στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τώρα, οι προϋποθέσεις. Υπάρχει μια διαδικασία για τις προϋποθέσεις για να αναθεωρούμε τις προϋποθέσεις. Κοιτάμε τις στρατιωτικές δυνατότητες χρειαζόμαστε για διάφορα σενάρια. Εντοπίζουμε ότι θέλουμε δυνατότητες κυβερνοάμυνας. χρειαζόμαστε κάποια ποσοτικά στοιχεία, νούμερα δηλαδή, ώστε να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, καθώς και ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή τα πρότυπα, η αλληλεπίδρασή τους κτλ. Για τις ασκήσεις, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να συνεισφέρουμε σε στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις Υπάρχει μια, ε, κάποια γυμνάσια, κάποιες ασκήσεις που τελείωσαν με τους Ισπανούς και ετοιμαζόμαστε για πολυμερείς τώρα ασκήσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Απάτσι. Ε, βάζουμε τις προϋποθέσεις και συνεργαζόμαστε με τους ανατοητούς συμμάχους για να δούμε τι διαδικασίες έχουμε για να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουμε και να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε και να υποφεληθούμε. Για την ανάπτυξη δυνατοτήτων ε, συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό, υποφελούμαστε ε, από την πραγματογνωμοσύνη του. Ε, μέσω από τις ειδικέ ομάδες που έχουν για τα κυβερνοθέματα αλλά και τις διαδικασίες ΠΕΣΚΟ. Επίσης, συνεισφέρουμε και συνεισφέρουμε στην κοινή κοινοποίηση της Κομισιόν και της επίσης Εξωτερικής Δράσης που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2017, ούτω ώστε να ενισχυθεί το θέμα της κυβερνοάμυνας και κυβερνοασφάλειας. Στην κοινή ανακοίνωση ίσως είδατε ότι ένα από τα παρτήματα ήταν ένα προσχέδιο που κοιτούσε το μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση κρίσεων. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητε ΚΠΑ συνάδουν με τις προϋποθέσεις για την υποβολή εκθέσεων ε, που βαραίνει τα θεσμικά όργανα. Αυτά. Θα σταματήσω και ακούω και τις ερωτήσεις αν έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριοι. Πολύ τεχνική παρουσίαση. Εξαιρετικά σημαντικό το θέμα. Σημαντικότατο για μας να είμαστε ενήμεροι για τις εξελίξεις. Κύριε Γκάλερ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη καταρχάς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, που με εμπόδισαν να έρθω νωρίτερα. Στο τέλος, στην τελευταία παρουσίαση, διαπίστωσα ότι ήταν σαν να είχα ξανακούσει αυτά που είπατε όσον αφορά τι δραστηριότητε παρακολούθηση. Απαιτήσει για παιδεία κατάτηση και ασκήσεις για την ασφάλεια. Παρόμοια διατύπωση είχαμε στην έκθεσή μας και ήμουν εισηγητή για την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της ΚΕΠΑ και θέλαμε να δημιουργήσουμε αντίσταση και αντοχή μέσω εκπαίδευση, μαθητείας κλπ. Και να αλλάξουμε το όλο τοπίο της εκπαίδευσης κατά σε θέματα ασφάλεια. Εσείς το προωθείτε ή υπάρχει φυσικό ενδιαφέρον από πλευράς κρατών μελών. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη. Τα κάτι πλευρά πιέζουν. Αυτά ακολουθούν αυτή η κινητηρια δυναμη τα κατι μελη πιεζουν αυτα ακολουθουν αυτη την κατευθυνση και συνεργάζεστε. Ή εσείς τους πρόχνετε. Ποιος παρακινεί, ποιος παρακινείται. Και το τοπίο εκπαίδευση και μαθητείας, τι σημαίνει. Ότι έχουμε ένα δίκτυο που λειτουργεί εθνικών κέντρων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και που συνεργάζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα εντατικά. Ευχαριστώ. Κλέρ, θες να πεις και εσύ κάτι. Ευχαριστώ όπως και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γκάλερ, ζητώ συγγνώμη πραγματικά που δεν ήμουν παρούσα για όλη την παρουσίασή σας. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να, τα, να μελετήσουμε ε, το θέμα και τις παρουσιάσεις. Έχω κάποιες προθεσμίες να τηρήσω και γι' αυτό ήμουν εκτός εθούσης. Τι είπατε ότι είχατε κάποιες επιθέσεις που έχουν διαπιστωθεί. Η εξωτερικής δράσης έχει σχετικά πληροφορίες. Ποιος κρύβεται πίσω τις επιθέσεις, ξέρουμε. Στο τέλος της παρουσιάσεως αναφερθήκατε στο δρομολογηθέν έργων, συνεργασία με άλλους οργανισμούς διερωτάς το ποιες διαδικασίες υφίστανται για ε, διαβίβαση πληροφοριών με τον ΝΑΤΟ. Ανταλλαγή πληροφοριών με τον ΝΑΤΟ. Η κατάσταση αλλάζει ραγδαία. Νέα τεχνολογία εφαρμόζεται. Υπάρχει τεχνογνωσία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπάρχει σχετικός μηχανισμός. Όχι μόνο με τον ΝΑΤΟ, αλλά και συνεργασία με άλλους τομείς. Τώρα για τους ορισμούς. Αν υπάρχει κάποιο επεισόδιο διαδικτυακό, υπάρχει κάποια κοινή προσέγγιση με τα κράτη-μέλη και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τι ορίζεται ως κυβερνοεπίθεση, περί τίνος πρόκειται. Και σχεδιασμό, σωστός. Κυβερνοάμυνα εκ των προτέρων, όχι σαν μέσο διορθωτικό. Σίγουρα θα τα καλύψατε αυτά, αλλά αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Η Κλέρ Μούντι, αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής. Η κυρία Άννα Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, πραγματικά συγκλονίστηκα με αυτά που μας είπατε. αν έχετε προχωρήσει στο στρατιωτικό τομέα μετά το 2012 και πήγατε από ένα στο 2,5 άτομα που ασκούν τα καθήκοντά τους, τι να πω. Να γελάσω, να κλάψω, ας κλάψω. Και δεν υπάρχει ολοκλήρωση, ενιαία προσέγγιση κυβερνοασφαλείας, κυβερνοαμήνης. Όταν ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε ε, απειλές, κατσαπλιάδες που μας επιτίθενται. Είναι απίστευτη η σπατάλη πόρων όταν δεν έχουμε καν πόρους. Και ελάχιστε επενδύσεις. Είναι κρίσιμο το θέμα. Αφορά τις αποστολές ΚΕΠΑ, τους γειτονές μας, τους στόχους μας. Θέλουμε ισχυρότερη κυβερνοασφάλεια και σχετική στατηγική άμυνα Ευχαριστώ που μας τα γνωστοποίησατε όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε πολλές ερωτήσεις και ας επευθύνουμε προς υπευθύνους. Εσείς υποφέρετε από τις συνέπειες και προσπαθείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε. Δεν φταίτε εσείς. Σε ποιο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας παράγων που εμπόδισε καλύτερη συνεργασία του τομέα του πολιτικού με το στατιωτικό και των σχετικών δομών. Σε ποιο βαθμό μόνιμο αρχηγείο θα έκανε την διαφορά για την ΚΕΠΑ. Σε ποιο βαθμό, όπως είπατε αναφέρετε την Ουκρανία. Η Ουκρανία προφανώς είναι η αποστολή που είναι πιο επιρρεπή στις κυβερνοεπιθέσεις. Σε ποιο βαθμό λέγω αυτό τι εικόνα που παρουσιάστηκε είναι πραγματική. Πώς αυτή η διαπίστωση δεν οδήγησε σε μεγαλύτερες επενδύσεις για τα απαραίτητος ε, αναγκαία. Σας ευχαριστώ που μας ενημερώσατε. Καλώς. Το τέλος των παρεμβάσεων από τους παρισταμένους συναδέλφους θα ζητήσω από τα μέλη του πάνελ να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών. Σας ζητώ συγγνώμη, διότι πρέπει να αποχωρήσω. Σας ζητήσω από την Κλέρ Μούντι να έρθει εδώ και να αναλάβει την προεδρία της υποεπιτροπής. Ας ακολουθηθεί η ίδια των απαντήσεων. Ο κύριος Χούμπερ και μετά ο κύριος Νιερ Παύλου. Ε, Θα ήθελα να προσθέσω λίγα σχόλια για την εκπαίδευση, κατάρτιση και ασκήσεις οπωσδήποτε υπάρχει υψηλός βαθμός ενημέρωσης τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται αλλά Μόλις τώρα αρχίζουμε να ξεκινάμε τέτοιες αποστολές, θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε αποσπασμένους ανθρώπους από τα κράτη-μέλη. Και υπάρχει το ίδιο πρόβλημα που έχουμε όλοι, ότι οι ειδικοί αυτοί είναι σπάνιοι. Οπότε υπάρχει και ζήτημα προσφοράς. και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εκπαίδευση και κατάρτιση και η θέληση να αυξήσουμε ακριβώς ε, τα επιχειρησιακά τμήματα στις αποστολές που θα παρέχουν αυτή την εκπαίδευση. Το κομμάτι δεν της εμπειρίας θα το αφήσω στον συναδελφό να κάνω, αλλά ένα σχόλιο τι είναι τόσο σημαντικό αυτό και γιατί πρέπει να γίνει τόσο νωρί. Τα πάντα κοστίζουν. Εάν υπάρχει μια αξιολόγηση κινδύνου που δείχνει ότι το επίπεδο προστασία επικοινωνιών και εγγράφων από κατσαπλιάδε ε, πρέπει να είναι ψηλό, ε, τότε έχουμε έναν παράγοντα κόστους που υπολογίζεται βεβαίως όταν ε, συζητάμε με τα κράτη-μέλη. Η προστασία επίσης των πληροφοριών, Η αρχιοθέτηση. Και επίσης ε, ε, την σημασία της. Τι άλλο. Το ερώτημά σας κυρία Γκόμες ε, για τη μόνιμη έδρα με το αρχηγείο αν θα έκανε καμία διαφορά. Κοιτάξτε, δύο χρόνια είμαι εγώ σε αυτή τη θέση μόλις. Τότε η ομάδα μας ήταν ε, ένας ε, ε, εθνικός εμπειρογνώμονας που ήταν δωρεάν για μας. Και τώρα έχω έξι άτομα και άλλες τρεις θέσεις στην διαδικασία πλήρωσης. Οπότε ήταν τεράστια η προσπάθεια και βεβαίως ε, έχουμε το κοινό αυτό κέντρο και την πλατφόρμα. Πέρσι, ε, τέλος του 2016, ε, έλαβα 7 θέσεις και το συμφώνησαν αυτό τα κράτη-μέλη πέρσι τον Δεκέμβριο και τώρα πληρώνονται άλλες 5 στον τομέα της επιμελητίας και της πληροφορικής. Στην πληροφορική, για να υπολογίσω, είναι 8 οι Πολύ σημαντικό αυτό. Και όλα αυτά βεβαίω, ε, δεν συνοδεύονται με μηδενικέ περικοπέ ε, στην πλευρά των αποστολών. Αν δούμε λοιπόν αναλογικά ε, σε σχέση με άλλα θεσμικά όργανα. Είμαστε πολύ χαμηλά. 2,4% του προσωπικού μα είναι στην πληροφορική, παρόμοιο επίπεδο με την ΕΕ. Δεν πρέπει να ομολογήσω όπου βεβαίω ε, σε διοικήσει όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στη Γραμματεία του Συμβουλίου είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό. Έχει γίνει όμως σημαντική προσπάθεια ε, και βεβαίως μία μόνιμη έδρα θα έκανε διαφορά. Ο δε επικεφαλής της, αντιπροσω... της ε, υπηρεσία πληροφορική τον, τον επισκέφτηκα, είπε είμαστε πέντε άτομα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε αν θέλουμε λοιπόν κάτι το σαφές ε, στη βαρύ υποδομή που να αντέχει σε ε, επιθέσεις χρειάζεται μια μονάδα Ακούσατε πως ε, στην στρατιωτική πλευρά υπάρχει η διεύθυνση πληροφορικής, ενώ εμείς έχουμε κομμάτι ενός τμήματος. Όλα όπως σας είπα σημειώνεται πρόοδος. Από τον έναν πήγαμε στους 8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης και κατάρτισης νομίζω το τονίσαμε ε, νομίζω ότι ωφελούμαστε από την αυξανόμενη ενημέρωση των 100 μελών. Τώρα, το ποιο ε, θίγει για κάτι τέτοιο ε, είναι από διάφορε κατευθύνσει. Εμείς, ας πούμε, στην ε, ομάδα ε, την στρατιωτική της εκπαίδευσης εισάγουμε τις διάφορες απαιτήσει, αλλά και η ΕΕΔ έχει κάποιες αρμοδιότητες ε, την πτυχή της εκπαίδευσης του προσωπικού, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δουλειάς τους. Και αυτά είναι βεβαίω και προς όφελος των κρατών μελών, οπότε είναι λίγο από όλα θα Είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι για να στήσουμε μια πλατφόρμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αξιολόγησης ε, που θα έχει φτάσει σε μια αρχική επιχειρησιακή φάση φέτος τον Σεπτέμβριο. Ένα θετικό μήνυμα αυτό νομίζω. Όσον αφορά το ευρύτερο τοπίο υπάρχουν αρκετοί πάροχοι τέτοια εκπαίδευση όμως το θέμα είναι τι προδιαγραφές έχει αυτή η εκπαίδευση. Θα επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι της αμοιβία αναγνώρισης. Χρειάζεται κάποια συγκριτική αξιολόγηση για να πούμε αν κάτι ε, επαρκεί ή όχι. Οπότε εντάξει είμαστε εκπαιδευμένοι άνθρωποι και μπορούμε νομίζω να κάνουμε μια αξιολόγηση για το τι σημαίνει αυτό. Ε, βεβαίως ε, από την πλευρά των πληροφοριών ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται συνεχώς και πρέπει να είμαστε σε επαφή με την ευρύτερη κοινότητα για να λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες. Και μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα όσον αφορά τον διαμοιρασμό πληροφοριών. Έχουμε λοιπόν την ε, ανταλλαγή πληροφοριών με τον ΝΑΤΟ, έχουμε τον οδικό χάρτη, κάποιες βασικές πληροφορίες που όλοι συμφωνούμε ότι μπορούμε να τις μοιραστούμε. Έχουμε λοιπόν το άτυπο επίπεδο για να γνωρίζουμε όλοι το τι κάνει ο καθένας. Όσον αφορά λοιπόν το μέγεθο τη ομάδα, είμαστε μικρή ομάδα, δρούμε στο στρατηγικό επίπεδο, υπάρχει αρκετό φόρτο εργασία και είναι κάτι το οποίο γίνεται εσωτερικά αυτή τη στιγμή στο στρατηγικό επιτελείο, στο στρατιωτικό μυστικό επιτελείο. Αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα βεβαίω που εμπλέκονται έργο αυτό και σημαντικό για μας είναι να βρούμε ακριβώς την αιτιολόγηση για τις αποστολές έτσι ώστε όταν αναπτύσσονται και ζητάνε χρήματα ή πόρους από τα κράτη-μέλη να είναι αιτιολογημένο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι ο ρόλος μας θα έλεγα για την κυβερνοασφάλεια σε σχέση με την κυβερνοάμυνα. Συνεργαζόμαστε με τους πολίτες συναδέλφους μας στο κοινό στρατηγείο και τη μονάδα συντονισμού και όταν αναπτυχθεί αυτό νομίζω ότι θα έχουμε πολλά ωφέλη στο μέλλον. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και με την ΕΕΔ, την πλευρά πολιτικής ασφαλείας. Ε, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα γιατί σαφώς αντιμετωπίζουμε κάποιες απειλές. Το άλλο θέμα για στρατιωτικό πολιτικά ζητήματα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, οπότε δεν θα το απαντήσω. Και απαντήθηκε νομίζω το ερώτημα για την ε, έδρα, το στρατηγείο μας. Σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας και για τις ε, παρουσιάσεις σας. θα είμαστε σε επαφή. Uh, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Α συμμαζευτούμε. Πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξή μα. Το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων και τη EDA. This item we και του, ελληνικού, του Ευρωπαϊκού Μυντικού Μηχανισμού. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ρότζαρ που είναι διευθυντής των Ευρωπαϊκών Συνεργειών και Καινοτομιών στον Ευρωπαϊκό Φορέα Άμυνας και είναι διευθυντής για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα ο άλλος συνάδελφος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση των αμυντικών προσπαθειών της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε είναι περίπλοκο θέμα. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικείμενη άμυνα και, και πάθα αποτελέσουν ε, κινητήριο δύναμη για συνεργασία για διάφορα σκηνοπραξίες αφορά του εξοπλισμού. Άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω προσπαθούν να αντιμετωπίσουν από διαφορετική οπτική γωνία το θέμα. Οπότε η σύσταση συνεταιριστικού οικονομικού μηχανισμού για οικονομική υποστήριξη ανάπτυξης στρατιωτική τεχνολογίας εστιαζομένη επί τεχνολογίας διπλής χρήσεως δείχνει τα ωφέλη εφάντας της συνεργασίας και την προθυμία που έχουν οι εμπορευόμενοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προχωρήσουν πραγματικά. Όμως, η αδίποτε φιλόδοξη πρόταση θα πρέπει να ακολουθείται από εξίσου φιλόδοξη υλοποίηση Γι' αυτό προσβλέπω στο να ακούσω τι έχουν να μας πούν οι φιλοξενούμενοι μας σχετικά με ποια συγκεκριμένα προγράμματα θέλουν να δρομολογήσουν αρχικά, πώς οι νέες διαδικασίες που συνδέονται με την ΠΕΣΚΟ, πώς θα κινηθούν και πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τις όσε προσπάθειες. Σε αυτή τη φάση θα ήταν κατάλληλο να δώσω το λόγο στον κύριο Ρότζο ε, για να μας εκφράσει την άποψή του και να μας κάνει την παρουσίασή του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Όχι. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκλησή σας στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο την κυρία Μούντι για την ε, πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά και τιμή ήρθα εδώ για να σας μιλήσω για τη συνεργασία ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως ξέρετε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Άμυνα ε, δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τον αμυντικό τους ε, μηχανισμό και δυνατότητε για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τι κρίσει και να υποστηρίξουν την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνα. Για 20 χρόνια η μείωση του αμυντικού προπολογισμού ήταν κάτι που αντιμετωπίζαμε συνεχώς η αμυντική βιομηχανία και οι ένοπλες δυνάμεις πάντα εξέφραν τις ανησυχίες τους για τον κίνδυνο που απορρέει από αυτή την τάση. Το 2015 η τράπεζα ε, έδωσε μεγαλύτερη σημασία στον τομέα αυτό και αντέστρεψε τις ε, δημοσιονομικές τάσεις. Ε, αλλαγή έγινε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Στρατηγικής από την ύπατη εκπρόσωπο ε, μέχρι την πρόσφατη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης όπως τη μόνιμη διαφθομένη συνεργασία που είναι η ΠΕΣΚΟ. Ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Μηχανισμός πάντα τόνιζε το εξής, ότι είναι σημασία να ξοδεύουμε αλλά καλύτερα οι, τα 27 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον οργανισμό ε, έχουν, ε, το, το, δεύτερο μεγαλύτερο προπολογισμό για αμυντικά θέματα με τι ΗΠΑ. Το θέμα δεν είναι το να ξοδεύουμε, αλλά το πώ θα ξοδεύουμε. Η συνεργασία, εναρμόνιση των προποθέσεων και παγίωση των ε, α, μεθόδων ε, για να αυξήσουμε την ποιότητα των δαπανών. Τον Δεκέμβριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Χαρισμό να δει πώς μπορεί να δώσει κίνητρα για οικονομική συνεργασία ε, στον αμυντικό τομέα. Ε, Παραδείγματος χάρη εξαιρέσεις ε, από φόρους για προγράμματα συνεργασίας, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επερδίσεων. Ε, για να υπάρξει καλύτερη διαρθρωμένη συνεργασία ανάμεσα στους, στην τράπεζα και τον οργανισμό, ε, υπογράφτηκα ένας, ένα μνημόνιο συνεννόησης από δύο επικεφαλείς των δύο οργανισμών. Πιστεύουμε στο τεράστιο δυναμικό αυτής της συνεργασίας για να αυξήσουμε την ποιότητα των δημοσίων απανών και να ε, αυξήσουμε και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών ε, με σεβασμό των πολιτικών των δύο οργανισμών. Το Μνημόνιο Συνεννόησης έβλεπε τέσσερα παραδοτέα. Καταρχάς την υποστήριξη μέσα στα πλαίσια της εντολής του κάθε συμμετέχοντα, της εφαρμογής των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών που συνεισφέρουν στην ε, ασφάλεια και άμυνα στο ύψος της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας, υποστήριξη στην ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας Ευρώπης, ανάπτυξη και συμμετοχή της τράπεζας στις ε, δραστηριότητες του οργανισμού, δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα στην τράπεζα και στον οργανισμό για να υπάρξουν συνέργειες και στήριξη προς το, τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών και ανταλλαγή πραγματογνωμοσύνης στο αμυντικό και οικονομικό τομέα. Ο οργανισμός και η τράπεζα συνεργάζονται δηλαδή για να εντοπίσουν ε, επενδυτικές ευκαιρίε για την τράπεζα. Το αποτέλεσμα θα είναι να βρεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση για προγράμματα τα οποία έχουν ε, προβλήματα χρηματοδότησης ή επενδυτικές ανάγκες και που έχουν όμως το δυναμικό να ενισχύσουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, του αμυντικού κλάδου. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε τους διάφορους φορείς της άμυνας στα κράτη-μέλη, ε, εμείς, ο οργανισμός μάλλον, ε, δίνουμε το, την ε, εμπειρογνωμοσύνη μας προς την τράπεζα, αλλά και ένα ειδικό εργαλείο, ε, ένα μηχανισμό συνεργατικής οικονομικής συνεργασίας, μια και οι δημοσιονομικές, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός των κρατών μελών αλλάζει, προσαρμόζουμε και το χαρτοφυλάκιό μας. Και εμείς, τα κράτη-μέλη, μπορεί να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο project, αλλά δεν είναι σε θέση, γιατί δεν έχουν τους πόρους, ε, αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν γιατί δεν έχουν τους πόρους. Η τράπεζα υπάρχει εκεί για να μην υπάρχουν τέτοιες χαμένες ευκαιρίες, δίνοντας τους οικονομικούς πόρους προς τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Παράλληλα, Βεβαίω, α με διορθώσει ο συνάδελφο από, από την τράπεζα. 80 εκατομμύρια δανείζονται από την τράπεζα. Ε, μερικά αμυντικά προγράμματα είναι πολύ μεγάλα. Ε, μιλάμε για εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια για την ανάγκη χρηματοδότησης. Ε, υποστηρίζει η τράπεζα τις ανάγκες των κρατών μελών Το CFM σχεδιάστηκε για να υποστηρίζουμε τη φάση δρομολόγησης συνεργατικών προγραμμάτων. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η συνεργασία επάσχει λόγω του ότι δεν έχουν οι διάφοροι εταίροι σε ένα πρόγραμμα τις ίδιες ε, οικονομικές δυνατότητες. Ε, γι' αυτό έχουμε καθυστερήσεις ε, στα προγράμματα και χάνουμε και πολλές ευκαιρίες κάποια προγράμματα να οδηγήσουν σε βιομηχανικά προϊόντα. Ε, τα κράτη-μέλη όμως, ε, χάρη σε εμάς, μπορούν να δείξουν τι, ενδιαφε... τους ενδιαφέρει, ε, ποια προγράμματα τους ενδιαφέρουν. υπάρχουν κοινέ προϋποθέσεις και αυτή είναι κρίσιμη φάση, ούτως ώστε να πετύχει συνεργασία. Ο, ο καθορισμός αυτός, ο ορισμός αυτός χρειάζεται χρόνο. αυτό μπορεί να, σημαίνει, μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη ίδιων αναγκών οικονομικών και οικονομικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Το σύστημα αυτό έχει και ένα δεύτερο πυλώνα που βασίζεται στη συνεργασία με την τράπεζα ε, ως ε, δανειτή, δανειστή. Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις τα προγράμματα, η τράπεζα θα διαπραγματευτεί με τα ενδιαφεροντα τη κράτη-μέλη ε, για να ξεκινήσει μια πιστοτική γραμμή για κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Οι μεταφραστές σας ζητούν να μιλάτε γαλλικά, λέει η ομιλήτρια. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σας καταλάβουν. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς, αλλά όχι για μένα, λέει ο Γάλλος ομιλητής. <laughs> Okay. Λύσω πιο αργά, αλλά στα αγγλικά. Ο σκοπός της ε, προσπάθειας αυτής της τράπεζας είναι ακριβώς να, ανοίξει, να δώσει μια πιστοτική γραμμή για κάθε συμμετέχον κράτος μέλος με ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο ποσό και ένα ε, προκαθορισμένο επιτόκιο. Σε αυτό το σενάριο, ο οργανισμός χρησιμοποιεί την ε, πραγματογνωμοσύνη του για να αξιολογήσει τα προγράμματα των κρατών μελών και τις μεθόδους για να δούμε ποια είναι η δυνατότητα να επιλεγούν ε, κάποια προγράμματα για χρηματοδότηση. Συζητάμε ακόμα με την τράπεζα και τα κρατημέλη τις λεπτομέρειες για το ρόλο της, του οργανισμού στη διαδικασία επικύρωσης των προγραμμάτων. Ειδικά δεδομένη της περιπλοκότητας και των διαφόρων αποχρώσεων της έννοιας της διπλής, ε, προϊόντων διπλής χρήσης και τεχνολογίας διπλής χρήσης, η τράπεζα δείχνει το ενδιαφέρον της για να αυξήσει την υποστήριξή της προς ε, την ατζέντα άμυνας και ασφάλειας στην πρωτοβουλία της Ευρώπης για την ασφάλεια και την άμυνα που παρουσιάστηκε. Το πλαίσιο αν μα ζητηθεί να το κάνουμε, μπορούμε να προσφέρουμε την πραγματογνωμοσύνη μα για να αξιολογήσουμε διάφορα προγράμματα ε, υποστηρίζοντας την τράπεζα. Ο οργανισμός κάνει μια ανάλυση για την πιθανή χρήση ενός τεχνολογικού στοιχείου, προϊόντος, ε, αξιολογούμε τον διτό χαρακτήρα, βλέπουμε μήπως έχει ε, βασικά στρατιωτικά χαρακτηριστικά αλλά και πιθανή πολιτική χρήση. Σε τι φάση είναι το κάθε project, το κάθε πρόγραμμα. Όσο πιο καθυστερεί, όσο πιο χαμηλά είναι η τεχνολογική εξέλιξη, όσο πιο υπολείπεται, τόσο πιο πολύς χρόνο χρειάζεται για να περάσει το προϊόν στη φάση υλοποίησης. Βλέπουμε αν ε, μόνο η αμυντική βιομηχανία είναι αποδέκτης του προϊόντος ή υπάρχουν πολύ, ένας ευρύτερος κύκλος χρηστών. Ο οργανισμός μέσω αυτών των δραστηριοτήτων και πολλών άλλων μπορεί να εντοπίσει ποια προγράμματα ή τμήματα των, τμήματα των προγραμμάτων είναι επιλέξιμα για την χρηματοδότηση της τράπεζας ο οργανισμός παίζει και το ρόλο του διευκολυντή, ετοιμάζει μορφότυπους για την συγκεκριμένη λειτουργία του CFM. Το βασικό αποτέλεσμα της ε, συμμετοχής της τράπεζας οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση και ευελιξία των συνεργατικών προγραμμάτων. Αυτό τελικά οδηγεί σε ακόμη περισσότερη συνεργασία, παγίωση και ενδυνάμωση της ασφάλειας των πολιτών. Φερρυπίν δεν είναι αποκλειστικό αυτό που λέω, κάποια project μπορούν να υποφεληθούν από την ε, δυνατότητα ε, χρηματοδότησης ε, χάρη στο CFM. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς για να είμαστε το συντομότερο δυνατό έτοιμοι. Πρέπει να τονίσω ότι η διαδικασία είναι συμπληρωματική με άλλες πρωτοβουλίες που είναι εξελίξει, εξελίξη. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, Φερπίν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει μια οικονομική εργαλειοθήκη για να προωθήσει τη συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Ο οργανισμός ε, συμμετέχει σε αυτές τις προσπάθειες. Όχι μόνο είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ε, που διερευνούν πιθανά εργαλεία, αλλά προσφέρει και την πραγματογνωμοσύνη του ε, από το 2014 προς τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, αμοιβαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην, στο Διοικητικό Συμβούλιο του CFM, ε, εξασφαλίζοντας ότι οι δύο τραπεί προχωρούν παράλληλα και με πλήρη διαφάνεια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το CFM μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε μια πρώτη φάση και πολύ αργότερα μπορεί να εσωματωθεί στην ευρύτερη εργαλειοθήκη εάν το επιθυμήσουν τα κράτη-μέλη. Συμπερασματικά, το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να σας ε, στείλω είναι το εξής. Πρώτον, ο οργανισμός δουλεύει προσφέροντας κίνητρα για συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Θέλουμε να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις και να τις δώσουμε στους ενδιαφερόμενους φορείς. Όλα τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν είναι εντελώς εθελοντικά. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν εάν θέλουν να συμμετάσχουν και δεύτερον, αργότερα, εάν θέλουν να ζητήσουν την υποστήριξη της τράπεζας. Θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να λάβουν, ή μάλλον τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν αυτή τη βοήθεια χάρη στα εργαλεία που έχουμε. Ε, υπάρχει εξορθολογισμός των ταπανών στους διάφορους τομείς, Υποστηρίζουμε την διαδικασία και σεβόμαστε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων της τράπεζας και τον τρόπο δανειοδότησης. Προς το παρόν λειτουργούμε στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής δανειοδότησης της τράπεζας. Εάν χρειαστεί να υπάρξουν τροποποίησεις της πολιτικής δανειοδότησης της τράπεζας, τόσο ώστε να υποστήριξουμε πολύ περισσότερα προγράμματα, τότε αυτό θα πρέπει να το εξετάσουν τα κράτη-μέλη και προφανώς όχι η ίδια η τράπεζα και θα το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Σε αυτή την φάση απλώς προσφέρουμε την πραγματογνωμοσύνη για αμυντικά θέματα ε, προς την τράπεζα, ε, προς το συμφέρον των διαφόρων φορέων των κρατών μελών. Επίσης, θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν τις αμυντικές δυνατότητές τους ε, με τη συνεργασία της Κομισιόν Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε για λεπτομέρειες και ερωτήσεις. Κύριε Μούντ, σας παρακαλώ εσείς. Madam Chair, members of Parliament. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται να ομιλήσει πρώτη επιτροπή. Χαιρόμεθα ιδιαίτερω για την ευκαιρία αυτή. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας το τι θα κάνουμε στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, εστιαζόμενοι επί της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Αν δεν σας πειράζει, επειδή περισσότεροι δεν γνωρίζετε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σύντομη επισκόπηση των εργασιών μας. Ah, um, e η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στόχος της χρηματοδότηση μακροπροθέσμων επενδύσεων σε όλη την Ένωση και μέσω εντολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βασίζεται από δύο θεσμού, την Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Το Ταμείο είναι στην διοκτησία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικών Τραπεζών ε, και, και κυρίως με κεφάλαια κινδύνου ασχολείται το Ταμείο και η Τράπεζα με τη δανειοδότηση. Είμαστε ένας από που δημιουργήθηκε το 58, άρα γιορτάζουμε, 60η επέτειος φέτος. Βασικός σκοπός, χρηματοδότηση για ανάπτυξη, για απασχόληξη και στήριξη της ανταγωνιστικότητας τα κράτη-μέλη είναι οι ιδιοκτήτε μα. Και τα 28 κράτη-μέλη είναι οι ιδιοκτήτε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα ποσοστά φαίνονται στη διαφάνεια. Όπω και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, ανήκουμε, είμαστε θεσμό που ανήκει στα κράτη-μέλη. Αυτό που ξέρουν ελάχιστοι. Είμαστε ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειοδότη και δανειολήπτης στον κόσμο μεγαλύτερη και την Παγκόσμια Τράπεζα καμιά φορά, σε κάποιες περιπτώσεις. Βασική δραστηριότητα αφορά τουλάχιστον 450 προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε όλο τον κόσμο, με ελάχιστε εξαιρέσει. Έδραμα στο Λουξεμβούργο. Έχουμε πολλά υποκαταστήματα και τοπικά γραφεία. Με ελάχιστου ανθρώπου εκεί. Είναι κεντρική η διοίκηση και γι' αυτό είμαστε πολύ αποτελεσματικοί έχουμε περίπου 3.500 ε, υπαλλήλους προσωπικό. Αυτά λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα. Αντικατοπτρίζει το τι έκανε μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Τι βλέπετε από την γραφική παράσταση. Συναρτήση του χρόνου. Μετά το 2001 έχουμε δανείσει 6 δις ευρώ σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε άμυνα, αεροδιάστημα, κυβερνασφάλεια. Αν κάποιο σα δείχνει από τράπεζα τέτοιο γράφημα, πρώτη ερώτηση είναι τι θέλει να μου πει αυτό όταν μου δείχνει το γράφημα. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι δεν το παρακολουθούμε συστηματικά το θέμα. Είμαστε νέοι στον τομέα, νέοι εισερχόμενοι. Από τις διακυμάνσεις τι βλέπετε όποτε υπήρξε κάποιο αίτημα από κάποια επιχείρηση για χρηματοδότηση, έρευνα και ανάπτυξη νέα τεχνολογία, εμπεριείχε κάποια στοιχεία διπλής χρήσεως, αλλά δεν ήταν ε, το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας αυτό. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια μπήκαν στη χρηματοδότηση καινοτομία και τα συναφή προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεω. Και η τρέχουσα χρηματοδότηση στα πλαίσια τη καινοτομία κατ' είναι 30, 13 δι ευρώ. Βλέπετε εδώ το συσχετισμό. Ήταν πολύ μικρό κομμάτι τη δανειοδότησή μα. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διερευνήσει δυνατότητες αυξήσεως της υποστηρίξεως στις πολιτικές ασφαλείας και άμυνας, κυρίως στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας και ανάπτυξης. Το Δεκέμβριο πέρσι, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλείας, που συναθρίζει τις δραστηριότητε της τραπέζης, την στήριξη που παρέχει προς τον τομέα της άμυνας και της ασφαλείας στην Ευρώπη. Θέλαμε να αυξήσουμε τη δανειοδότηση και δεσμευτήκαμε να παράσχουμε 6 δις ευρώ χρηματοδοτήσεως την επόμενη τριετία. Το ίδιο ποσό που δώσαμε από το 2001 μέχρι τώρα θα το δώσουμε σε τρία χρόνια. Ε, σημαντική αλλαγή και νέα στοχοθέτηση των δραστηριοτήτων μας. Τι θα κάνουμε. Θα σας δείξω τώρα. Έχουμε τα τμήματα εκείνα που πιστεύουμε ότι εντός της εντολής μας και των πολιτικών μας μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Έχουμε τέσσερις τομείς. Ο πρώτος, πολιτική έρευνα και ανάπτυξη στον πολιτικό τομέα. Έρευνα και ανάπτυξη για τεχνολογίες ασφαλείας. Δεύτερον, τεχνολογίες διτής χρήσεως, στατιωτική συνιστόσα, πολιτική συνιστόσα, τρίτος τομέας, κυβερνοασφάλεια και βιοάμυνα, τέταρτο τμήμα, υποδομές ασφαλείας, ό,τι σχετίζεται με τις μεγάλες υποδομές, στρατηγικές υποδομές στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα γίνουν εντός του πλαισίου πολιτικών της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων. Κάτι που καθορίστηκε μαζί με την δυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέσω καταλόγου αποκλειστικών δραστηριοτήτων που καθορίστηκε που εδράζονται επί στατιωτικού τομέα πυρομαχικών εξοπλισμού αστυνόμευσης Εκεί μάλλον δεν μπορούμε να επενδύσουμε στους τομείς. Διότι η πολιτική Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ευθυγραμμίστηκε με άλλου διεθνείς χρηματοστηρικούς οργανισμούς όπως Φερρυπίνη Παγκόσμια Τράπεζα. Δεύτερον, δεσμευόμεθα από αυστηρότατες αρχές για το περιβάλλον και οι κοινωνικές πτυχές συμμορφωνόμαστε. Υπάρχει σαφής πολιτική περί εξορισμού υποθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να αποκαλύψει κάθε χρηματοδότηση, κάθε ε, επένδυση που πραγματοποιεί. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε τη νέα πρωτοβουλία περί ασφαλείας με τους περιορισμούς που προανέφερα. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συζητήσαμε για κάποιο χρονικό διάστημα το θέμα και δοκιμάστηκε το θέμα και σε συζητήσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνης και έχουμε την πεποίθηση ότι τηρώντας με αυστηρότητα τους περιορισμούς παράλληλα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σειρά επενδύσεων για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μέχρι 6 δις ευρώ μπορούμε να δανειοδοτήσουμε την επόμενη τριετία. Αυτό που κάναμε ήδη είναι μία-δύο χρηματοδοτήσεις που θέλω να σας αναφέρω, δεν σας πειράζει, ξεκινώντας με τα κεφάλαια κινδύνου. Έχουμε κινηθεί όσον αφορά τις επενδύσεις κινδύνου για θέματα που άπτονται της αμήνης, αλλά κυρίως για τεχνολογίες ε, διπλής χρήσεως. Αυτό επιτυχάνεται κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Δεύτερο παράδειγμα. Η Τάρμα, η ε, αμυντική βιομηχανία από τη Δανία, δώσαμε ένα δάνειο 30 εκατομμύρια. Σε αυτή την ε, δανέζικη εταιρεία για να αναπτύξει εφαρμογές για τον πολιτικό τομέα, για τεχνολογίες ραντάρ. Δάνειο που υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ή Ρίστον παρόδο είναι μια εταιρεία που είναι νέος πελάτης της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, αλλά δεν είχαμε χρηματοδοτήσει πριν αυτή την επιχείρηση, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και αυτή και άλλες παρόμοιες εταιρείες όπως η ΤΑΜΑ και στο μέλλον στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας στην ασφάλεια άλλη εταιρεία. Η Άβιο, Ιταλική ε, εταιρεία αεροναυπηγικής και διαστήματος, χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη νέων κινητήρων ε, πυράβλων από το Βρασάβιο. Και πάλι δάνειο που υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Άρα εντό των εγγυήσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τέλο, εξίσου η βαβαρική Nordic. Παραπλανά ο τίτλος είναι δανέζικη εταιρεία αυτή. Είναι από τους μεγαλύτερους ε, ερευνητές και αναπτύσσουν εμβόλια. Και ο μεγαλύτερος πελάτης κατά το παρελθόν ήταν το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα είμαστε στη δεύτερη χρηματοδότηση, εξετάζουμε δεύτερη χρηματοδότηση της εταιρεία αυτής. Υπάρχει μεγάλο ε, ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό. Όχι μόνο των αμυντικών δυνάμεων, αλλά και των πολιτών. Αυτή είναι μια σφαιρική εικόνα, μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων μας. Τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέλλον. Σχεδιάζουμε τη χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα. Και εδώ μπαίνω στη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνας δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα και την αμυντική βιομηχανία που είναι από τους δικαιούχους της χρηματοδοτήσεως αλλά έχουμε και το δημόσιο τομέα για την δημόσια έρευνα και ανάπτυξη και κάποιες επενδύσεις για υποδομές που απαιτούνται. Ξανά, στα πλαίσια της διπλής χρήσεως και των συναφών τεχνολογιών για την ασφάλεια που αποκλείουν το, τους βασικούς τομείς του στρατού και της αστυνομίας. Κάποιους τομείς αναφέρω. Το Μνημόνιο Συνεννόησης με την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνης θεσμοθετεί κατά κάποιο τρόπο τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης. Βασικός σκοπός αυτού είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά η τεχνογνωσία που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμήνης και δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον ε, τομέα της αμήνης και της ασφαλείας είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια της ε, αμήνης πρέπει να βασιστούμε για την τεχνική αξιολόγηση των σχετικών επενδύσεων επί της τεχνογνωσίας, τεχνογνωσίας συγγνώμη, της του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης, κυρίως επί της ως κατά πόσο κάποια τεχνολογία είναι διπλής χρήσεως ή όχι. Ο λόγος γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάποια έτη, δεκαετίες χρηματοδοτήσεως νέων τεχνολογιών, αλλά όχι σε αυτόν τον τομέα και δεν έχουμε τους εμπειρογνώμονες ούτε την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την αξιολόγηση εντός του φορέα μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερω λοιπόν που μπορούμε να βασιστούμε επί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης για την αξιολόγηση των τεχνολογιών αυτών. Αναφερθήκατε ήδη προηγουμένως στα περισσότερα από αυτά που βλέπετε εδώ. Δεν θα τα αναφέρω για να ξεκονομήσω χρόνο. Κλείνοντας, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απεφάσισε να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοδότηση και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ασφαλείας και Αμήνης στους σχετικούς τομείς. Θα παράσχουμε χρηματοδότηση όποτε κριθεί αναγκαίο, κυρίως όσον αφορά τον όγκο στον ιδιωτικό τομέα, στις αλυσίδες ε, εφοδιασμού, κυρίως επί μικρομεσαίων και μεσαίων προς μεγάλες επιχειρήσεις θα και επί του δημόσιου τομέα, με βασικό στόχο τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνη στα πλαίσια τη προσπάθεια για την άμυνα, την Ευρωπαϊκή, και των επικειμένων συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο τη Άμυνα. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω τον λόγο στους ε, συναδέλφους. Ο Μιχαήλ Κάλερ πρώτος. Ναι. Θα μιλήσω γερμανικά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενική εικόνα που μας δώσατε και καλό θα ήταν να μας ε, τα στείλετε αυτά και γραπτός. Εγώ θεωρούσα ότι όταν προσεχώς στο πλαίσιο ε, και πά τα κράτη-μέλη θέλουν ε, να χρηματοδοτήσουν ένα έργο, τότε θα έχουμε μια τέτοια συμφωνία όπως αυτή που κάνατε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αποφευχθεί μια κατάσταση που θα οδηγούσε στο ότι θα έχουμε διαφορετικούς κύκλους ε, Χρηματοδότηση και σχεδιασμού των Υπουργείων Αμήνη που θα καθιστούν την κατάσταση αδύνατη. Βεβαίω αυτά είναι εθνική υπόθεση το πόσα λεφτά έχει κανείς φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου. Και βεβαίω ε, τα έργα τα οποία σχεδιάζει κανείς. Και αν πει κάποιος ότι θα εξοικονομήσουμε λεφτά κάνοντας κάποια πράγματα μαζί, και τα βρίσκει όλα αυτά λογικά. Έρχεται ο Υπουργό Οικονομικών ή όποιο είναι αρμόδιο για τα οικονομικά στο Υπουργείο Αμήνη και λέει κύριε Υπουργέ, δυστυχώς ε, περιθώριο έχουμε σε 3, 4, 5 χρόνια και δεν μπορεί να δώσει ο Υπουργός το πράσινο φως. Και ε, τότε, κατά την δική μου την άποψη, το ιδεώδες είναι να υπάρχει η δυνατότητα να πει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, μέχρι να μπορέσετε να πληρώσετε σε τρία χρόνια, ξέρω εγώ, είτε μιλάμε για έρευνα είτε για προμήθεια, για τα τρία χρόνια θα πληρώσουμε εμείς. Τα γράφουμε δηλαδή και μας τα χρωστάτε και όταν ε, ολοκληρωθεί το έργο θα μπορούν να το εκμεταλλευτούν όλοι. Εάν έχω καταλάβει τώρα καλά, ο τομέας για τον οποίο ισχύει αυτό το οποίο παρουσιάσατε γραπτός έχει ως έξις ε, ε, η αμυντική έρευνα δεν ε, περιλαμβάνεται εδώ ή δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή θα με ενδιαφέρει αυτό στον τομέα της έρευνας και στον τομέα της άμυνας εάν δεν είναι διπλής χρήσης. Και το άλλο, όταν μιλάμε όντω για την προμήθεια καθ' αυτή η οποία ε, αποκλείεται ας πούμε να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για τρία χρόνια για να αποκτηθούν από κοινού κάποια οχήματα. Έτσι είναι ή έχω καταλάβει λάθος. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην συνάδελφο την κυρία Λέζινγκ. Ναι, ναι. Δεν θα μιλήσω κι εγώ αγγλικά για να μην υποφέρουν οι διερμηνείς. Στα γερμανικά λοιπόν λέμε ότι με αυτό που χαίρεται ο ένας θυμώνει ο άλλος. Δηλαδή αυτό το οποίο εκνευρίζει τον κύριο Γκάλερ μπορεί να χαροποιεί την δική μου ομάδα. Γιατί βεβαίως εμείς δεν υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση στρατιωτικών έργων και ε, ότι έχω καταλάβει και εγώ και ο κύριος ε, Γκάλερ θα ήθελα να επιμείνω στο εξής ε, το πώς το ορίζετε εσείς αυτό δηλαδή μιλάτε για τομείς, κλειδιά στρατού και αστυνομίας, αλλά αποκλείονται οι επενδύσεις στον δημόσιο τομέα. Αυτό είναι θετικό. Επίσης, και αυτό με τα εμβόλια, δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο συνδέει κανείς με Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία ή πρόγραμμα έρευνας. Και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε παρά τους ε, περιορισμούς. Αυτό είναι και το δικό μου το ερώτημα και θεωρώ ότι πράγματι είναι μια σημαντική προοπτική και υπάρχει και η ιστοσελίδα σας την οποία μελέτησα όπου λέτε ότι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε έργα τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Ο κύριος Ροζέ είπε σαφώς ότι μιλάμε για τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων του αισθήματο της ασφάλειας ε, κτλ. Καλά. Ε, καλό είναι το ότι τα λέει καθαρά και ανοιχτά. Αλλά εδώ προκύπτει μια αντίφαση, έτσι. Υπάρχουν ε, αμερικανικές έρευνες που ξεκαθαρίζουν ότι οι επενδύσεις στον τομέα της άμυνας τελικά συνεισφέρουν λιγότερο και στην ε, απασχόληση σε σχέση με άλλη έρευνα. Γιατί λέμε ότι ένα δολάριο στην έρευνα ε, αποδίδει περισσότερο στην πολιτική έρευνα από ό,τι στον τομέα των εξοπλισμών. Οπότε και αυτό δεν ταιριάζει με αυτά τα οποία μας λέτε και θα ήθελα κατόπιν να μάθω σε ποιο βαθμό είναι δημόσιο αυτό το μνημόνιο, στην αντίληψη, αν μπορούμε να το δούμε. Και μιλήσατε επίσης για διαφάνεια θα έχουμε κάποιες ε, πληροφορίες για το τι θα, γίνει, τι θα γίνουν αυτές οι πιστώσεις και ποιες πιστώσεις θα έχετε. Μια που είμαι πρόεδρος θα κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες από τις οποίες προκύπτουν από τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Αναφέρατε κύριος Τιρελ. Και προφανώς όσο χαμηλότερο το επίπεδο τόσο λιγότερη είναι η... ο βαθμός της Οπότε αναφέρατε και τους περιορισμούς της ε, πολιτικής. Και αναρωτιέμαι ποιοι θα είναι αυτοί. Τι εννοείται δηλαδή. γιατί η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι. Επίσης, είμαι περίεργη για αυτό το οποίο είπατε για τα εμβόλια και πώς ε, ταιριάζει με τις αμυντικές δαπάνες. Και επίσης προφανώς ένα από τα κίνητα για την στήριξη ανάπτυξης ε, της αμυντικής χρηματοδότησης αφορούσε ακριβώς την αποφυγή του να κάνουμε τέτοια πράγματα δύο φορές. Και βεβαίως το τι στοιχεία υπάρχουν ε, σε σχέση με αυτό. Αν υπάρχουν, βέβαια μπορεί να μην υπάρχουν. Ευχαριστώ και αναμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ξεκινώντας με το τι εστί άμυνα και ασφάλεια και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κύριε Γκάλερ, για να απαντήσω. Σαφώς η προμήθεια όπλων, οπλικής τεχνολογίας, οπλικών συστημάτων ε, δεν θα είναι δυνατή. Απαγορεύεται. Σαφώς αποκλείεται. Σε γενικές γραμμές η προμήθεια στρατιωτικού υλικού είναι απίθανο να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση εκτός εάν ε, δεν είναι καθαρά στρατιωτική. Παραδείγματο χάρη υποστηρίζουμε τον εξυγχρονισμό στρατώνων δηλαδή η ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν είναι καθ' αυτό στρατιωτικές επενδύσεις, αλλά χρειάζονται. και κάποια άλλη τομείς π.χ. κάποια ανακαίνιση κτίριων και εγκαταστάσεων. Ο κύριος στόχος μας όμως είναι η έρευνα και η τεχνολογία και εξετάζουμε πολύ προσεκτικά επίπεδα TL όπου θεωρούμε ότι μέχρι το επίπεδο 4 μπορούμε να είμαστε ε, αρκετά σίγουροι ότι υπάρχει δυνατότητα διπλής χρήσης σε όλες αυτές τις τεχνολογίες. Σε κάποιους τομείς μπορούμε να φτάσουμε και στο επίπεδο 6. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό κατά περίπτωση. Και ο λόγος είναι ότι όποτε μιλάμε με την αμυντική βιομηχανία βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης ε, της τεχνολογίας είναι πολιτικό, μη στρατιωτικό. Οπότε, η προσαρμογή ε, πολιτικών τεχνολογιών στον στρατιωτικό τομέα, στηρίζοντας λοιπόν ε, την πολιτική έρευνα και ανάπτυξη, υποστηρίζουμε και ανάπτυξη αμυντικών εφαρμογών. Σκεφτείτε παραδείγματος χάρη το προφανές ε, του τομέα της πληροφορικής. Ε, όλα είναι εκεί πέρα πολιτικός ε, τομέας. Υπάρχει τεράστια ανάγκη κυβερνόμενας και έχει μείνει πίσω η Ευρώπη και ακριβώ βλέπουμε πως αυτό αφορά και προμήθειες κυβερνοασφαλείας από τον δημόσιο τομέα. Ένα άλλο θέμα είναι τα υλικά. Η έρευνα επί των υλικών είναι ε, κατά κύριο λόγο πολιτική έρευνα, μη στρατιωτική. Αυτά λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και ο λόγος για τον οποίο ε, εξετάζει η αμυντική βιομηχανία όλες αυτές τις εφαρμογές είναι ότι γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες επενδύσεις που χρειάζονται δεν θα γίνουν ποτέ από τον δημόσιο τομέα για την άμυνα. Έχουμε λοιπόν πολύ χαμηλές αμυντικές δαπάνες, οπότε χρειάζονται αυτές οι συνέργειες ή επειδή υπάρχει τεράστια πολιτική αγορά για αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να βρουν πολλές εφαρμογές για αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε κατά την άποψή μας καθαρά στρατιωτικές τεχνολογίες είναι ελάχιστες. Και αν είναι καθαρά στρατιωτικές τεχνολογίες δεν τις χρηματοδοτούμε. Και εκεί πέρα βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας για να μας πει ακριβώς ποιος είναι ο βαθμός αλληλεπικάλυψης μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Για να απαντήσω λοιπόν και στην κυρία Λέζινγκ, θεωρούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος τομέας όπου η τράπεζά μας θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες μας. Όσον αφορά τον πολλαπλασιαστή και αν υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και τις δουλειές. Ναι, θεωρούμε ναι. Ένας από τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές που έχουμε είναι στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, μακροπρόθεσμα. Οπότε είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν στηρίζει μόνο τον τομέα της άμυνας ε, όπως καθορίζεται στενά, αλλά υπάρχουν σαφώς επιδράσεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σε σχέση με το ερώτημά σας για τον εμβολιασμό, Προσπάθησα να το εξηγήσω στην περίπτωση της Berry ε, Nordic, η οποία ιδρύθηκε σε ένα πανεπιστήμιο και είχε μόνο έναν πελάτη. Έναν πελάτη επί 10 χρόνια. Και δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήγε σε αυτήν την εταιρεία. 100% χρηματοδοτούμενη από τον ιδιωτικό τομέα. Είχαν αποτελέσματα της έρευνας και πήγαν στην παραγωγή και μόνο όταν πάτησαν γεράτα στα πόδια τους όσον αφορά τις κρηματικές ροές άρχισαν τα, ε, την ανάπτυξη εμβολίων ε, μη στρατιωτικών πολιτικών. Ναι, για να φέρω έναν τομέα μόνο. Παραδείγματο χάρη ε, όλα αυτά τα εμβόλια της ανεμοβλογιάς. Προέκυψαν από αυτήν την εταιρεία. της ευλογίας, με συγχωρείτε. Και αυτό σχετίζεται με την ε, άμυνα και την ασφάλεια. Και θα ωφεληθεί βεβαίω και ο πολιτικός τομέας. Διαφάνεια. Εμάς μας δεσμεύει ο κανονισμός του άρχους για να αποκαλύπτουμε ό,τι είναι δυνατόν, ειδικά σε σχέση με το περιβάλλον και τα κοινωνικά ζητήματα. δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ε, εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες γιατί βασιζόμαστε και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, σταθμίζοντας τα συμφέροντα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε ιδιωτικές εταιρείε όταν μιλάμε για ευαίσθητα εμπορικά μυστικά δεν τα αποκαλύπτουμε μέχρι πλέον να μην είναι ευαίσθητα μυστικά. Όσον αφορά το μνημόνιο, δεν είμαι 100% σίγουρος για το αν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το εμπιστευτικό για την ανηλεπικάλυψη. Βεβαίω ο στόχος είναι να αποφύγουμε ακριβώς την ανηλεπικάλυψη και να ωφεληθούμε από την συνεργασία. Η έρευνα και η ανάπτυξη δηλαδή στον τομέα της άμυνας ε, που γίνεται από όλα τα κράτη μαζί οπότε να μην γίνονται πολλές φορές τέτοια πράγματα και να είναι καλύτερες οι δαπάνες και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων οπωσδήποτε στηρίζει αυτή την προσπάθεια αλλά μπορείτε να πείτε κι εσείς περισσότερα από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γκούναρ κάλυψε τα περισσότερα. Να συμπληρώσω κάποια στοιχεία. Το θέμα της επικάλυψης. Να έχετε υπόψη ότι η αφετηρία όλου του εγχειρήματο από πλευρά δική μα, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνη, είναι να δώσουμε κίνητρα όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα τη αμήνη. Να δώσουμε λοιπόν κίνητρα στα κράτη-μέλη να ενώσουν τι δυνάμει τους σε συνεργατικά προγράμματα αντί να κινούνται ξεχωριστά και να επαναλαμβάνονται οι προσπάθειες. Για μας όλες αυτές οι εξελίξεις, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επενδύσεων και η δημιουργία του CFM οδηγούν στη χορήγηση κινήτων οικονομικών για τη συνεργασία. Επίσης, μία επικάλυψη με τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως σας είπα, Επικρατεί πλήρη διαφάνεια, συνεργαζόμαστε με του συνεργάτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουμε στι δικέ συνεδριάσει, συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του CFM και όλο και περισσότερο αισθάνομαι ότι το CFM είναι πρόδρομο των μελλοντικών εξελίξεων όσον αφορά την εργαλειοθήκη ε, του Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμήνης. Λοιπόν, είναι καλό πρώτα απ' όλα να δοκιμάσουμε τις αρχές και αυτά τα μορφότυπα πριν να, μορφότυπους μάλλον πριν δαπανηθούν, ε, δαπανηθούν χρήματα. Τώρα, για τις τεχνολογίες και τους τομείς που καλύπτονται από το CFM και από τη συνεργασία ανάμεσα στον οργανισμό και στην τράπεζα, θα ήθελα να τονίσω ότι στο CFM, έτσι όπως είναι σχεδιασμένο σήμερα, υπάρχουν δύο σκέλη ένα δικυβερνητικό και ένα που το υποστηρίζει η τράπεζα. Στο πρώτο σκέλος μιλάμε για δάνεια. Με δόσεις, με δόσεις ε, μεταξύ των κρατών μελών. Και τι καλύπτει αυτό το σκέλος, ε, τα αναφέρει το άρθρο 5 της ε, απόφασης ε, του οργανισμού. Ε, αποστολές ε, δυναμικού έρευνας και τεχνολογίας, υποστήριξη στην ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογία κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα προγράμματα μπορούν να καλυφθούν. Mm. Αλλά μιλάμε για διακυβερνητικό σκέλος μεταξύ των κρατών Το δεύτερο σκέλος το οποίο ε, εμπλέκεται η τράπεζα, η τράπεζα, εδώ έχουμε διαφορετική κατάσταση. Θα πρέπει να σεβαστούμε εδώ την πολιτική δαδειοδότηση της τράπεζας. Ε, ενώ ο οργανισμός μπορεί να έχει έναν σύμβουλο που, που τον δανείζει στην τράπεζα και αξιολογεί τη φύση ενός προγράμματος, ελέγχει ότι το πρόγραμμα, ας πούμε, είναι πρόγραμμα διπλής χρήσης, για προϊόντα διπλής χρήσης. Ξέρετε ότι υπάρχει μια προ... διαμόρφωση προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού. Ε, βλέπουμε τις νέες τάσεις. Ακριβώς. Όλοι και περισσότεροι τομεί προτεραιότητα είναι τομεί διπλή χρήση και είναι στα όρια μεταξύ ασφάλεια και άμυνα. Ε, δόθηκαν πολλά παραδείγματα, ενέργεια, κυβερνοχώρος, υλικά, ε, ηλεκτρονική, ηλεκτρονικά στοιχεία. συστήματα εξοπλισμού, ε, ηλεκτρονικά συστήματα εξοπλισμού αεροπλάνων κτλ. Όλα αυτά έχουν όλο και περισσότερο διπλή χρήση, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Δηλαδή, στην πολιτική αντιοδότηση της τράπεζας, το 70 ή 80% των όσων εντοπίζουμε ως τεχνολογικές προτεραιότητες για την άμυνα είναι, οδηγούν σε προϊόντα διπλής χρήσης. Σε ό,τι αφορά το είδος των προγραμμάτων που θεωρούμε ότι μπορεί να προταθούν από τα κράτη-μέλη και για τα δύο σκέλη του CFM. Εκεί υπάρχει μια πλειάδα. Δεν θέλω να περιοριστώ στο TRL. Mm. Mm. Όσο χαμηλότερο είναι το TRL, τόσο μεγαλύτερη διπλή χρήση. Μπορεί σε επίπεδο ITRL να έχει πραγματικά προϊόντα διπλή χρήση. Οι προτάσει που περιμένουμε από τα κράτη-μέλη είναι διαφορετικής φύση. Προβλέπουμε κάποιες προτάσεις που αφορούν τα παραδοσιακά προγράμματα γιατί για κάθε ευρώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τα κράτη-μέλη. Μερικές φορές ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν μπλοκάρει ε, τον προϋπολογισμό για φέτος, ε, κάποια άλλα το έχουν αφήσει για του χρόνου. Στην περίπτωση λοιπόν ε, αυτή, ε, το CFM μπορεί να εξασφαλίσει ε, δανειοδοτικό συγχρονισμό για να ξεπεράσουμε τα δημοσιονομικά μπλοκαρίσματα. Έχουμε κάποιες αρχικές επαφές με τα κράτη-μέλη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό ε, συνεργατικής χρηματοδότησης για μεγάλα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη θέλω τώρα τον ε, εξοπλισμό μου, αλλά δεν έχω τον προϋπολογισμό ή θα τον έχω σε δύο χρόνια, ας πούμε. Μπορείς να με συνδράμεις, ας πούμε, ε, να μου δώσει μια βραχυπρόθεσμη λύση και το CFM μπορεί. Πολλές φορές στις ερωτήσει και στις παρουσιάσεις η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία ακούστηκε και αναφέρθηκε. Φαντάζομαι ότι μερικά από τα αμοιβαία προγράμματα ΠΕΣΚΟ θα μπορούσαν να υποφεληθούν από τη στήριξη του CFM, ούτως ώστε να δοθεί γρήγορη πίστοση, γιατί κάποια προγράμματα μπορεί να είναι πολύ νέα και τα κρατημέλη να δυσκολεύονται να βρουν την απαραίτητη χρηματοδότηση που είναι στο ύψος των φιλοδοξιών. Περιμένουμε ε, το τέλος του χρόνου για να οριστικοποιήσουμε τις διευθετήσεις για το CFM με τα κράτη-μέλη και να τσεκάρουμε το σύστημα αυτό ε, για να αποδείξουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα την πραγματική προσθέμενη αξία της συνεργατικής οικονομικής διαχείρισης του CFM. Καλύφθηκα νομίζω διάφορες ερωτήσεις έτσι, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, την πολιτική διαφάνειας. υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί μόνο για τα εμπορικά μυστικά, για τα εμπορικά απόρριτα. Περιορισμός της διαφάνειας λοιπόν. Συμπερασματικά το CFM είναι τμήμα μιας δέσμης νέων εργαλείων που έχουμε αναπτύξει πρόσφατα στα πλαίσια της νέας αμυντικής πολιτικής προσπάθειας και πλαισίου και θέλουμε με συγκεκριμένα επιτυχή παραδείγματα να πείσουμε τους Υπουργούς Άμυνας για να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα. Γιατί άλλοι υπουργοί είναι πολύ πιο συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους οικονομικά εργαλεία από τους πολύ πιο συνηθισμένους Υπουργούς Άμυνας. Γι' αυτό λοιπόν ε, προσπαθούμε όλοι μαζί για να τους δείξουμε ε, ότι είναι προς το συμφέρον τους να χρησιμοποιήσουν το CFM και είμαι σίγουρος ότι οι Υπουργοί Άμυνα θα ενδιαφερθούν πολύ περισσότερο στο μέλλον, ειδικά όταν έχουν κάποια προγράμματα έτοιμου παράδοτα για να τα προτείνουν και να τα υποβάλουν επιτάπητος. Ευχαριστώ. Και για την προηγούμενη παρουσίαση και τις διεξοδικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. θα δούμε παρόμοια θέματα σε μελλοντικέ συζητήσεις. Ήταν ενημερωτική η συνεδρίαση και εκτιμούμε πραγματικά το ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας να δώσετε τα στοιχεία σας. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Οπότε, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι καθήκον μου να σας ενημερώσω ότι η αυρενή συνεδρίαση ξεκινά στις 8.30 Ελπίζω να σας δω όλους πρωί-πρωί. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι.